Non, non, non, non, non. Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir les travaux. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να αρχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σας ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι της Επιτροπής Προϋπολογισμών, διότι σήμερα το πρωί είχαμε μια συνάντηση που κράτησε περισσότερο από ό,τι υπολογιζόταν, συνάντηση των συντονιστών, γιατί υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες σε σχέση με το προσχέδιο συμπληρωματικού διορθωτικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου φτάσαμε σε μια συμφωνία μεταξύ συντονιστών ως προς την επίλυση αυτού του τεχνικού προβλήματος. Θα μας απασχολήσει μετά από την ακρόαση από τις 11 και η ψηφοφορία για τον διορθωτικό προϋπολογισμό θα γίνει από τις 11 και μετά και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στο φάκελό σας θα προσθεθούν και νέες τροπολογίες που θα μας υποβάλει ο εισηγητής και θα μας επεξηγήσει αργότερα. Άμεσα έχουμε μια άλλη ψηφοφορία. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την ετήσια έκθεση 2008 ως προς την ΚΕΠΑ. Η κυρία Νάινσκι είναι η συγγήτρια. ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη μας παρουσίασε χτες την έκθεση και μαζί του θα συνεργαστούμε για την ψηφοφορία. Εάν λοιπόν είσαστε έτοιμοι, σας προτείνω να πάρετε τον κατάλογο ψηφοφοριών ως προς την έκθεση Νέισκη, στην παράγραφο 1 υπάρχει η τροπολογία 1 του κύριου Γκουαλτιέρη. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. 3-4. J'avais une mauvaise influence sur Bon. Euh, Αποχές. Καμία αποχή υπέρ εγκρίνεται. Στην παράγραφο 2, τροπολογία 2 της κυρίας Μπέρτμαν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές, καμία αποχή. Να συγχαρούμε την κυρία Βέρτμαν. Στην παράγραφο 8, τροπολογία 3 του κυρίου Γκουαλτιέρη. Υπέρ. Κατά. Αποχές Καμία αποχή, μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Ένας κατά. Στην παράγραφο 9 έχουμε την τροπολογία 4. Γουαλτιέρι Μπέγκε. Υπέρ. Κατά. 2 κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε τώρα την ε, έκθεση γνωμοδότης όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά ένας κατά αποχές μία αποχή. Σας ευχαριστώ. Άρα η έκθεση εγκρίνεται και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκουαλτιέρη. Περνάμε τώρα στο σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης. ως προς την κατάσταση στην Αϊτή μετά την τραγωδία του σεισμού. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε επίγουσες αποφάσεις που έχουν και οικονομικές επιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εγγράψει πιστώσεις στον προπολογισμό του 2006 μέχρι ενό ορισμένου ορίου. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, αυτή την τραγωδία και τις οικονομικές και ανθρώπινες συνέπειες, θα υπάρξει μία σημαντική χρηματοδοτική κινητοποίηση, άρα θα πρέπει να προβούμε σε αυτή την ακρόαση. Ο κύριος Ματσερβίση είναι Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και ο κύριος Τσάγκελ, Διευθυντής στην ΕΚΟ. Euh, ε, έχουμε καλέσει και εκπροσώπους από την ΑΦΕΤ και την Επιτροπή Ανάπτυξης για να προβούμε σε αυτή την ακρόαση. Ο κύριος Ματσαβής έχει το λόγο. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Θα ήθελα όμως να σας πω πού βρισκόμαστε και να σας δώσω και τις πρώτες απαντήσεις της Επιτροπής. Καταρχήν η κατάσταση στην ε, IT. Ο ε, ε, αρμόδιος επίτροπος παρευρέθηκε στην IT μαζί μου και με τον Πίτερ Ζάγκελ την προηγούμενη εβδομάδα για να δούμε πώς έχει η κατάσταση και να συντονιστούμε για να συντονιστούμε με τους άλλους εταίρους. Η κατάσταση αφορά μία ε, τραγωδία. Το Πόρο Πρένς έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερός και υπάρχουν πολλοί άστεγοι μέσα στην ίδια την πόλη. Πρόκειται για ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση παράλληλα. Θα πρέπει να πούμε ότι δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα σε αυτή την πτυχή, αλλά βρεθήκαμε σε μια χώρα όπου η αξιοπρέπεια των ανθρώπων ε, είναι πολύ υψηλή, δηλαδή μας έκανε εντύπωση πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις δυσκολίες, πώς οργανώνουν ξανά τη ζωή τους, την απαρχή μιας ζωής και δραστηριοποιούνται για να προβούν σε μία αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μόνο η σκοτεινή πλευρά, ε, προσπαθούν οι ίδιοι οι κάτοικοι της ΑΕΤΗΣ να αναλάβουν την κατάσταση και δεν δίνεται δημοσιότητα στο γεγονός ότι η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη, πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Όταν δεν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχουν μεγάλες εντάσεις. Όταν αντίθετα ε, υπάρχουν ε, τακτικές προμήθειες Βλέπουμε ότι οι κάτοικοι της ΑΕΤΙΣ ε, μπαίνουν στη σειρά για να πάρουν νερό από μία δεξαμενή ή για να λάβουν τρόφιμα. Ακόμα και η παρουσία της αστυνομίας και των στρατιωτικών υπάρχει, υπάρχει και προσδίδεται νέα διάσταση σε αυτήν. Έχουμε να ζήσουμε μία τραγωδία αλλά ε, δεν δίνεται δημοσιότητα σε όλες τις πτυχές, ιδιαίτερα στην ένταση. Ως προς την, τον συντονισμό της διεθνούς βοήθειας, αυτό είναι ουσιώδες ζήτημα, διότι προωθούμε ανθρωπιστική και κατεπίγουσα βοήθεια συνεχώς και κατά αποδοτικό τρόπο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει άμεσος συντονισμός έτσι ώστε να μην υπάρχει ο τρέχον ανταγωνισμός και να υπάρχει συντονισμός με τα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρξε άμεση επέμβαση από πολλούς εταίρους, ιδιαίτερα από πλευράς Καναδών και Ήπα, για την ανθρωπιστική βοήθεια με την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Θα περάσουμε όμως σε, έναν άμεσο συντονισμό των Ηνωμένων Εθνών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και για την αναγνώριση των διαφόρων καταβλισμών για να μπορέσουμε να τους προμηθεύουμε με είδη και ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε να προωθήσουμε ένα διάλογο με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την επόμενη φάση. Οι δημόσιες αρχές δηλαδή να μπορέσουν να αναλάβουν την ανοικοδόμηση γύρω από το πόρο Πρένς. Υπάρχει και το υπόλοιπο της ΑΕΤΙΣ που δεν υπολείπεται σε ανάγκες ανοικοδόμησης. Έτσι λοιπόν θα προωθήσουμε τις πρώτες μας δράσεις και επικεντρωνόμαστε σε τρία επίπεδα. Καταρχήν την κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ο Πίτερ Βάγγελ θα σας μιλήσει για αυτή. Η δεύτερη πτυχή είναι η κατεπίγουσα μη ανθρωπιστική βοήθεια. Αποτέλεσε αντικείμενο ε, συζητήσεων με τον ε, Επίτροπο ε, Ντεγκούχτ και τον ε, Πρόεδρο Μπελερίβ για να δούμε πώς το κράτος της ΑΕΤΙΣ θα αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του. Δηλαδή να λειτουργήσει ως κυβέρνηση και να παρέχει υπηρεσίες. Έχει σημασία λοιπόν η ανοικοδόμηση του κράτους. Περνάμε λοιπόν σε αυτήν την πρώτη φάση κατεπίγουσας μη ανθρωπιστικής βοήθειας. Από πλευράς πολιτικής δέσμευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για 100 εκατομμύρια ευρώ πρωτίστως, τα οποία θα είναι διαθέσιμα άμεσα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την μη ανθρωπιστική βοήθεια. Το τρίτο επίπεδο αφορά την ανοικοδόμηση καθεαυτή. Η ανοικοδόμηση θα γίνει στα πλαίσια μιας διάσκεψης που θα συγκληθεί το Μάρτιο που προετοιμάστηκε στο Μοντρεάλ την προηγούμενη Δευτέρα. Για τις δύο αυτές φάσεις υπάρχουν 100 εκατομμύρια για τις άμεσες μη ανθρωπιστικές ανάγκες και 200 εκατομμύρια για την ανοικοδόμηση. Πρόκειται για ενδεικτικά ποσά, τα οποία βασίζονται στα μέσα που διαθέτουμε. Ιδιαίτερα ως προς τα 100 εκατομμύρια. Τα 100 εκατομμύρια βασίζονται σε δύο χρηματοδοτικές πηγές. Η πρώτη είναι ο προϋπολογισμός, δηλαδή το μέσο σταθερότητας, το οποίο θα κινητοποιηθεί για 20 εκατομμύρια ευρώ και η δεύτερη συνιστόσα είναι το Food Facility, το οποίο ήταν έτοιμο προς δαπάνηση και θα χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη φάση μη ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από το 10ο έτα ή από το 1ο έτα. Ως προς το 10ο έτα, για το Vulnerability Flex, προτείναμε τις ε, δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή αυτό το safety net, το οποίο είχαμε ήδη ορίσει, 30 δηλαδή εκατομμύριων. Έχουμε το Β5 και 6 εκατομμύρια, τα οποία θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν άμεσα, και δύο προγράμματα του 1 του ΕΤΑ που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ε, ποιότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 5 και κάτι εκατομμύρια και ένα πρόγραμμα ανάκαμψης 33 εκατομμυρίων και κάτι. Αυτά αποφασίστηκαν, θα επαναχρησιμοποιηθούν, άρα φτάνουμε σε 100 εκατομμύρια, ένα ποσό που διαθέτουμε άμεσα και που μπορούμε να προωθήσουμε είτε εντός προπολογισμού είτε με βάση το ΕΤΑ σε συμφωνία με τις αρχές της ΑΙΤΙΣ. Γι' αυτό άρχισε και ο διάλογος με την κυβέρνηση. Συνεργαζόμαστε για να καταλήξουν σε, μια, ε, σε ένα νέο προσανατολισμό αυτών των ποσών. Την Κυριακή θα γίνει μία συνάντηση στην ΑΕΤ με, και με δικούς μας εμπειρογνώμονες σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη για να δούμε ποιες είναι οι κατά προτεραιότητα ανάγκες για αυτή τη φάση ανοικοδόμησης του κράτους. Δηλαδή, δεν να φτάσουμε σε ένα διοικητικό, να ανοικοδομήσουμε ένα διοικητικό κέντρο έτσι ώστε η κυβέρνηση να ορίσει τις προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες του κράτους. Τα 200 εκατομμύρια για την ανοικοδόμηση αφορούν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπόλοιπου φακέλου του 10ου ΕΤΑ με βάση τις ανάγκες που αφορούν την ανοικοδόμηση. Και εδώ θα συζητήσουμε με τους εταίρους και θα λάβουμε τις αποφάσεις με βάση τις τρέχουσες διαδικασίες για να αλλάξουμε τη ε, διαδικασία των ενδεικτικών προγραμμάτων εάν ε, ενδείκνεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή είναι και η εισήγησή μου. Ο κύριος euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για τι συμβαίνει επί τόπου σήμερα. Τώρα είχαμε τη γενικότερη εικόνα που μας την παρουσίασε σωστά ο Στέφανο. Ε, θεωρούμε ότι είναι ήπια η κατάσταση ήρεμη αλλά ασταθής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο αριθμός των αστέγων υπερβαίνει κατά πάσα πιθανότητα τις 250.000 για το Πόχτο Πχάνς, έτσι δεν μιλώ για τις υπόλοιπες πόλεις, γιατί προστίθενται άλλα αριθμητικά στοιχεία για τις άλλες πόλεις ε, είναι άστεγοι σε καταβλισμούς, ε, σε, στο δρόμο ε, και εκτίθενται στο, στις καιρικές συνθήκες. Προς το παρόν δεν βρέχει, οπότε όλα βαίνουν αισίως, αλλά αν αρχίσει να βρέχει τότε θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε οι αρχές της ΑΕΤ θα πρέπει ταχύτατα να βρουν κέντρα στέγασης ούτω ώστε η ανθρωπιστική οικογένεια στην ΠΟΕΤΣ να εγκατασταθεί και να προλιάνει το έδαφος ούτω ώστε να δούμε ποιες υγειονομικές ε, καταστάσεις, ε, εγκαταστάσεις υγειονομική περίθαλψης θα εγκαταστήσουμε και πρέπει αυτή η απόφαση να ληφθεί ταχύτατα. Όπως γνωρίζετε από ανθρωπιστικής πλευράς, ε, η Επιτροπή έχει ήδη κινητοποιήσει 30 εκατομμύρια ευρώ βάσει των προτύπων των δικών μας και ξέρω ότι εσείς χειρίζεστε ε, πολύ μεγαλύτερα ποσά, ε, αυτό το ποσό είναι πακτολός ε, και έχει τρεις συνιστώσεις. Πρώτον, πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας που ήδη τρέχει επί τόπου έτσι, και υπερβαίνει κατά τι το 20 εκατομμύρια για το 2009-2010 γιατί για την ΑΕΤ είχαμε τους κυκλώνες πέρσι ε, που, ε, και που οδήγησαν σε πολυάριθμους αστέγους και μεγάλες ζημιές αλλά είναι και ασθενές το κράτος, έχει διαρθρωτικά προβλήματα και έχει ε, οξύ ανθρωπιστικό πρόβλημα, υποσυτισμός, έλλειψη πόσιμου νερού, ούτως ή άλλως εδώ και καιρό λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας οπότε 8 εκατομμύρια χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Μετά το σεισμό το ανώτατο που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε 24 ώρες είναι 30 εκατομμύρια. Να σας, πω, να σας δώσω κάποια παραδείγματα, έτσι για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Τι κάνουμε με αυτά τα λεφτά. Ε, από τα 3 εκατομμύρια συγγνώμη δώσαμε ένα τμήμα στους ε, γιατρούς του κόσμου που έχουν ε, μέσα στο πανεπιστημιακό πανεπιστήμιο μία ε, μονάδα περίθαλψης ε, ε, και θα ε, νοσηλευθούν 15.000 άτομα περίπου. Τώρα κάτι άλλο που δεν είναι σημαντικό από οικονομική πλευρά αλλά έχει θεμελιώδη σημασία. Εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με την Telecom χωρί σύνορα, μια ε, μη κυβερνητική οργάνωση που έχει κάνει δύο πολύ βασικά πράγματα για την οργάνωση τη ανθρωπιστική βοήθεια στο αεροδρόμιο έχουν οργανώσει τη σύνδεση στο διαδίκτυο, έτσι, ούτως ώστε όλοι να μπορέσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με εμάς. Επίσης, τηλέφωνα στην πόλη, ε, ούτως ώστε οι πληγέντες να έχουν τρία λεπτά στη διάθεσή τους ε, για να τηλεφωνήσουν σε όποιον επιλέξουν για να τους ενημερώσουν για την κατάσταση της οικογένειάς τους. 60.000 ε, ευρώ είναι το κόστος, έτσι για να έχετε και μια ιδέα. Ε, επίσης, και στην πτυχή της πολιτικής προστασίας και στην ε, πτυχή της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, δίνουμε πόσιμο νερό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ε, να κάνω και άλλη μια παρατήρηση για το ανθρωπιστικό κομμάτι. Ε, η ρήψη από αέρος ε, της βοήθειας ε, δεν είναι η λύση που επιλέγουμε. Να σας εξηγήσω γιατί, έτσι. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η ρήψη από αέρος είναι η έσχατη, η εσχατότατη λύση όταν δεν μπορούμε να έχουμε αλλιώ πρόσβαση. Έτσι, αν δεν έχει προετοιμαστεί σωστά η επιχείρηση δε, ε, τραυματίζονται κάποιοι γιατί δεν ξέρουν πού θα πέσουν τα αγαθά. Ε, επίσης, Καταλαβαίνετε μια σύγχυση ακατανόμαστη έτσι, όταν προσπαθούν όλοι να ανοίξουν τα πακέτα. Δεν είναι ότι πρέπει να το απαγορεύσουμε, αλλά το χρησιμοποιούμε ως έσχατη λύση ε, και σε αστικές ζώνες όπως το Πόρτο Πράνς ε, αντενδείκνεται πλήρως η λύση, όπως είπε και ο συνάδελφος. Έτσι. Ε, και στο Πόρτο Πράνς έχουν ξεκινήσει κάπως οι ντόπιες δραστηριότητες, οι, λαϊκές κτλ. Και υπάρχουν πολλοί στην ουρά και περιμένουν να πάρουν τα προϊόντα με τη σειρά του. Αυτά. Τώρα, από πλευράς ε, προϋπολογισμού, ε, δύο στοιχεία. Όταν προγραμματίζουμε τα 800 εκατομμύρια της ΓΔ ΕΚΟ στις αρχές του 2010, το 80% ε, το προγραμματίζουμε για τις μεγάλες κρίσεις. Έτσι, Κονγκό, Τσάντ, Νταρφούρ, Αφγανιστάν, Εκεί πάει το 80%. Επίση, στα προπαρασκευαστικά μέτρα για τι φυσικέ καταστροφέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, το πιο πλέον σημαντικό ε, είναι να πούμε στου ανθρώπου τι πρέπει να κάνουν σε ένα πρώτο στάδιο και στη συνέχεια να κοινοποιήσουμε τι απαιτούμενε πληροφορίε. Οπότε, τον Ιανουάριο, στι αρχέ ε, ε, του έτους αρχίζουμε με 160 εκατομμύρια και πλέον που δεν έχουν διοχετευθεί και από παίρνουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για την ΑΕΤ προκειμένου. Γιατί το αναφέρω, γιατί αυτά τα 20% μας επιτρέπουν, θα έλεγα, ε, να καλύψουμε επαρκώς ε, μια συνηθισμένη χρονιά, έτσι, με τους κυκλώνες και τις φυσικές καταστροφές, πολλές και διάφορες. Δεν έρχομαι για να σας ζητήσω λεφτά εδώ σήμερα. Από τα 160 εκατομμύρια, πάνω από 20 ήδη έχουν ναι, αναλωθεί και ε, ε, να κάνω και μια χοντρική εκτίμηση, έτσι, ε, θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε τις ανάγκες για ένα δίμηνο περίπου. Όταν λοιπόν φτάσουμε στα κέντρα στέγασης και στους καταβλισμούς, έτσι, θα χρειαστεί επέκταση του σχεδίου προϋπολογισμού. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα αριθμητικό στοιχείο, έτσι, είναι πολύ νωρίς και είναι άσκοπο. Θα υπάρξει μια αποστολή αξιολόγηση των αναγκών και επί τη βάση της αξιολόγησης θα είμαστε πλέον σε θέση να σας δώσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεύτερον, ε, μία δυσκολία που δεν είναι τραγική και, εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε λύση εν τέλει. Ε, ξέρετε ότι ε, υπάρχει ένας ενθουσιασμός τώρα να καταστούν διαθέσιμοι πόροι από διαφόρους και από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και στη δική μας υπηρεσία, όμως, δεν έχουμε μηχανισμό ώστε να συλλέξουμε αυτά τα κονδύλια αυτούς τους πόρους. Δεν θα βρούμε λύση σήμερα ή αύριο, έτσι δεν το λέω για αυτό, αλλά καλό θα ήταν να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση. Με ποιο τρόπο θα καταστεί αυτό δυνατό, ε, διότι στο ενδιάμεσο διάστημα ε, οι αρχές ε, των κρατών μελών που έχουν πόρους, που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν διότι δεν έχουν προσωπικό, θα τις διαβάσουν στα Ηνωμένα Έθνη, όχι ότι έχουμε πρόβλημα. Ε, όμως για να προβάλλουμε ε, την ε, ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό θα ήταν να το εξετάσουμε για να ανοίξουμε και έναν άλλο διάβλο αν θέλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά για αυτή την περιγραφή που ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ε, ήταν ακριβής περιγραφή της κατάστασης και των προσπαθειών που ήδη έχουν γίνει. Ο εισηγητής του προϋπολογισμού 2010 θα ήθελε το λόγο τώρα, σε αυτό το στάδιο, κύριε Σούριαν. Ε, όχι, από ό,τι φαίνεται. Όχι, όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Ο Γέραν Φάρμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ακριβή παρουσίαση του θέματος που προσέφερε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αλλά έχω ορισμένες ερωτήσεις. Πρώτα, ορισμένες γενικές ερωτήσεις. Ίσως είναι κάπως πρόημο για να αξιολογήσει κανείς το τι έχει επιτευθεί, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε. Θεωρείτε ότι έχουμε την ικανότητα ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι τέτοια που να επιτρέψει ταχεία λήψη αποφάσεων διαβάζουμε στον τύπο ότι ασκείται πολύ κριτική κατά ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας λέγοντας ότι η ανταπόκρισή της υπήρξε αργή, ασυντόνιστη. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θεωρείτε εσείς ότι είναι αλήθεια. Και επίσης η συνολική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για το προφίλ της Ένωσης. Εκτός από τα 330 εκατομμύρια απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί πόροι που προήλθαν απευθείας από τις χώρες μέλη. Μπορείτε να μας δώσετε μια συνολική εικόνα του τι πράττουν Ένωση και μέλη και πώς γίνεται ο συντονισμός μεταξύ ενώσεως και μελών. Θυμούμε προπενταετίας με την ε, θεομηνία του τσουνάμι είχε υπάρξει σημαντική κριτική λόγω έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χωρών μελών σε ό,τι αφορά τι δυνατότητε μεταφορών κλπ. Ε, είδατε εσεί κάποια βελτίωση. Εν τέλει σχετικά με τα ποσά. Από αυτά που είπατε έως τώρα δεν μπορείτε να εξεύρετε τους απαραίτητους πόρους μέσα στον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Προβλέπετε ανάγκη νέων πόρων στο μέλλον που θα σημάνουν νέες αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και που ενδεχομένως θα έχουν επιπτώσεις σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού και μπορείτε σήμερα να πείτε κάτι το οποίο θα έχει σχέση με τους επόμενους μήνες. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Μπέγκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Γιώραν Φέρμ σχετικά με ένα σημαντικό θέμα το οποίο διαρκώς εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη αν θέλετε όταν αναλύουμε την αντιμετώπιση από πλευρά μα διαφόρων κρίσεων και όταν αναζητούμε τρόπους καλύτερου συντονισμού ε, παγκοσμίω και ε, κυρίως να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων και μη κρατικών οργανώσεων καλύτερο συντονισμός και Επομένως, βελτίωση και μεγαλύτερος επαγγελματισμός στην ανταπόκριση της κρίσης. Γνωρίζοντας βέβαια ότι οι θεομηνίες τέτοιου εύρους, τέτοιου μεγέθους ασφαλώς πάντοτε θα ε, καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ελλείμματα διότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι 100% προετοιμασμένος σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση που απαιτείται μετά από μια τέτοια θεομηνία. Τον Μάρτιο ακούσαμε ότι θα γίνει διάσκεψη δωρητών και ότι ακόμα θα χρειαστεί να εκτιμηθούν οι ανάγκες και επίσης το τι θα πρέπει να πράξει ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη τώρα εάν προ της διασκέψεως δωρητών θα συνομιλήσει με τις κοινοβουλευτικέ επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω έπραξε και η κυρία Φεραίρο Βάλτνερ παλαιότερα για την βοήθεια προ την Παλαιστίνη και ε, άλλα σχετικά. Για να δούμε και πώ θα διασφαλίσουμε τι διαδικασίε του προπολογισμού, ώστε να μην χρειαστεί ξανά να κάνουμε τέτοιες, τέτοιες ακροβασίες όπως κάναμε με την Food Facility. Είναι σημαντικό εφόσον προχωρήσουμε σε αυτήν την διάσκεψη δωρητών να μπορούμε να πούμε όχι ότι υπάρχουν προκαταρκτικές συμφωνίες αλλά ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράγματα τα οποία δεν θα είναι και μονομερή αλλά θα έχουν ήδη καλυφθεί από, ποια, από κάποιες πρώτες συζητήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπω ότι και από την Food Facility προβλέπεται 5,8 εκατομμύρια. Ακούω τώρα από τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι εν ώψη της καταστάσεως αυτής θα χρειαστεί ενδεχομένως να λαμβάνουν επιστηστική βοήθεια μέχρι 2 εκατομμύρια άνθρωποι για ένα έτος. Διεθνή επιστηστική βοήθεια. Εδώ τίθεται το ερώτημα τι γίνεται τώρα με την ε, εφαρμογή της Food Facility που είχαμε εγκρίνει και που τώρα συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι πόροι ή έχουν διατεθεί ήδη, έχει δηλαδή σχεδιαστεί η διάθεσή τους. Πρόκειται βεβαίω πρώτα για το νερό, τα τρόφιμα και τη φροντίδα της υγείας που αυτά πρέπει να διασφαλιστούν. Υπάρχουν από την Food Facility άλλοι διαθέσιμοι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τους επόμενους μήνες υπέρ της IT. Σας ευχαριστώ. Μπόκρος. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πολλοί μίλησαν για την ανάγκη συντονισμού. Ρωτώ πώς συντονίζεται το έργο διασώσεως με τους Αμερικανούς. Έχω την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί έχουν αναλάβει τα ηνία του εγχειρήματο όχι μόνο γεωγραφικής γυτνιάσεως αλλά και λόγω στρατιωτικής ισχύω που διαθέτουν στην περιοχή αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν να μας εξηγήσουν τι γίνεται, ποια συνεργασία υπάρχει μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Και το άλλο και τι είναι κάπως νωρίς ακόμη. Βλέπω εδώ οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση, που σημαίνει ότι ήδη αρχίζετε να σκέπτεστε και πέραν της ανθρωπιστικής βοήθειας πώς να αναζωογονήσετε την οικονομία. Κάτι βέβαια το οποίο θα είναι σημαντικό, κρίσιμο για την επιβίωση της αιτινής οικονομίας. Αν μπορείτε να αναπτύξετε κάτι σχετικά. Κατά τα άλλα, με έχετε εντυπωσιάσει πραγματικά με τα όσα κάνετε. η Σιδονία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα έχετε καταφέρει όλοι βλέποντας την ε, τραγωδία της ΑΕΤΙΣ ε, έχουμε κατά νου το τι θα μπορέσει να συμβεί από τώρα και στο εξή, διότι οι κάτοικοι της ΑΕΤΙΣ θα χρειαστούν ε, βοήθεια για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Γνωρίζουμε τα πόσα υπομένουν αυτός ο λαός. Και θα ήθελα να αποβάλω μια ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα προωθήσει αυτή την εργασία, πώς θα την προγραμματίσει αυτό το έργο δηλαδή να χορηγήσουμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν αυτά τα ποσά μετά από τη διάσκεψη των δωρητών. Εστιάζουμε την προσοχή σε δύο θέματα. Πώς εκτελείται η ανθρωπιστική βοήθεια, με τι ρυθμό, επιτοπίως πώς μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν, να δοθούν αυτά τα μέσα, πώς συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη ή με τις ε, μη κυβερνητικές που βρίσκονται επί τόπου. Πώς μπορούμε να χορηγήσουμε αυτή τη βοήθεια. Υπάρχει μία αποστολή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω κατά πόσο όμως επαρκεί για τις ανάγκες είναι επαρκές μέσων για να χορηγήσει όλη αυτή τη βοήθεια επί επιτοπίως. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά αυτό που προείπαν και μερικοί. Πώς έχουν οι δημοσιονομικές ανάγκες πώς μπορούν να οργανωθούν μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τη φετινή χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Μπορείτε να το αποτιμήσετε, να μας πείτε ποιες θα είναι οι ανάγκες για τα επόμενα έτη. Και αν όχι τώρα, πότε θα έχουμε τα πρώτη, τις πρώτες ενδείξεις για τις ανάγκες σε αυτό το τομέα. Ε, Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ Ευχαριστώ να προσθέσω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις για τα θέματα συντονισμού. Μία ερώτηση για την κατεπίγουσα βοήθεια των πρώτων ε, ημερών, θέμα πολυδοσκόπησης, έτσι. Πώς αντιδράτε στην προσπάθεια του Συμβουλίου για τη συγκρότηση δύναμης τύπου ΕΦΑΣΤ για να συντονιστεί η κατεπίγουσα βοήθεια των πρώτων ημερών, έτσι, ε, για να σωθούν ζωές, ανθρώπινες ζωές τις πρώτες ώρες και τις πρώτες ημέρες μετά από μια τέτοια τραγωδία. Ε, σε αντιδιαστολή με τις ε, σκόρπιες προσπάθειες ε, από διάφορες χώρες που στέλνουν σωστικά συνεργεία με κάποια ταξία σύγχυση γιατί είναι και χρονικό θέμα, θέμα ωρών, θέμα ημερών. Ο συντονισμός δεν μπορεί να χωλένει έτσι και να υποφέρει από την παραμικρή καθυστέρηση. Μια ευρωπαϊκή δύναμη τύπου Fast λοιπόν, πώς αντιδράτε σε αυτή την ιδέα και έχετε και εκτιμήσεις δημοσιονομικές ακριβώς τι θα συνεπάγεται αυτό η απόφαση συγκρότηση δύναμη ανεξάρτητα από την ανασυγκρότηση, τη διάσκεψη των δωρητών κτλ. Έτσι, χωριστά από όλα αυτά. Ευχαριστώ, με Ιζαμπέλο, κύριος ε, Λαβίρ. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση για να κατανοήσω πώς ε, ορισμένες παρεμβάσεις του προϋπολογισμού είναι χρήσιμες για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Μέσα στα πλαίσια του Leading 2 έχουμε ένα ποσό για ανθρωπιστική βοήθεια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε για άμεση παρέμβαση ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους. Άρα ίσως στο μέλλον θα έπρεπε να επαναπρογραμματιστούν για άλλους σκοπούς. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο οι πόροι που προορίζονται για αυτούς τους στόχους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή όχι ή θα χρησιμοποιηθούν ε, για άλλους σκοπούς πέρα από, τα προϊόντα από αυτό το πόσο που έχουμε για τα προϊόντα της αγοράς. Κύριε Βέρτμαν. Μιλήσατε συγκεκριμένα για δύο μήνες όπου ακόμη μπορεί κανείς να επιτύχει πολλά πράγματα. Μετά το δίμηνο αυτό, τι θα γίνει. Στους δύο αυτούς μήνες μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχουμε τόσα πολλά πράγματα ώστε η επιβίωση της χώρας αυτής να είναι δεδομένη ή πώς θα βοηθήσουμε τους Αίτινους περισσότερο. Επίσης θέλουμε να βοηθήσουμε είμαι βέβαια αρχάρια εδώ και δεν γνωρίζω καλά τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού αλλά δεν θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ένα ειδικό κονδύλιο για να το έχουμε έτοιμο ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις ε, ακροβασίες που είπε πριν κάποιος ώστε να έχουμε χρήματα όταν προκύψει κάποια θεομηνία. Η κυρία Χάουκ διευθύνει τώρα τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Λάζλο Σούριαν. Ευχαριστώ. Πρώτα θέλω να πω ότι δεν ήταν απλώς καλό το ότι έχουμε τώρα μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει, ένα καλό ενσταντανέ, έχουμε και κάτι άλλο θετικό. Είναι καλό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται με ειδικά προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Γιατί στο παρελθόν χρειάστηκε να δημιουργήσουμε αυτήν την πηγή χρηματοδότησης όταν είχε πια γίνει κάτι, όταν είχε συμβεί μια θεομηνία. Νομίζω ότι έχουμε τώρα μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη προσέγγιση βασισμένη στα βήματα που έχουμε ήδη κάνει. Μιλούμε για πάνω από 313 εκατομμύρια από διάφορες πηγές. που μπορούν να διατεθούν. Μιλούμε δηλαδή για μια προσέγγιση πιο όρθη που δεν θα σημάνει και η υπερβολική επιβάλληση του προπολογισμού για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εκτός αυτών των επιχειρημάτων, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας φροντίζοντας ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορούμε να δρούμε και να αντιδρούμε με τρόπο εύκαμπτο και ε, ταχύ. Δεν προσπαθώ να κάνω καμία κριτική για τα βήματα που έχουμε ήδη κάνει. Υποστηρίζω το την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της και νομίζω ότι ε, καλά τα έχει κάνει. Στην Ολομέλεια μιλήσαμε ήδη για την τραγωδία της ΑΕΤΗΣ και θελήσαμε να κάνουμε μια χειρονομία. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις βαρύτητα της επιπτώσεις αυτής της θεομηνίας και θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους που νομίζω ότι εν τέλει θα αποδειχθούν επαρκείς. Άρα θα έπρεπε να δώσουμε πλήρη υποστήριξη στην προσέγγιση της Επιτροπής και να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω προσπάθειες εάν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο. Και βέβαια χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι είναι πολύ σημαντικό εάν πρόκειται να κάνουμε μεταφορές πιστώσεων εάν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε άλλο εγώ βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας ως εισηγητής για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο μας με το σωστό τρόπο στο διεθνές προσκήνιο αποδεικνύοντας ότι σεβόμαστε τις ευθύνες μας και προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται σύμφωνοι με τις δυνατότητές μας. Ο Ρομπέρτο που μόλις κατέφτασε γιατί βεβαίως κατά τα άλλα είχαμε εξαντλήσει τον κατάλογο των αγορητών. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω μια θετική σκέψη για την κινητοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω μία ανησυχία ως προς την ε, ε, βραδύτητα της Επίτροπης κατά την προηγούμενη θητεία της κατά την προηγούμενη θητεία της ως προς την προστασία, πολιτική προστασία, την έκθεση Μπαρνιέ, είχαμε την έκθεση Μπαρνιέ, τη, τα δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟΝ το προηγούμενο Σεπτέμβριο. Όλα αυτά συνέκλειναν υπέρ της ενίσχυσης των Monitor Formation Center θα πρέπει να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στις συνθήκες, δηλαδή να προστατεύουμε τους πολίτες. Βλέπουμε όμως ότι όλα αυτά αποδυναμώνουν τη δυνατότητα συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επιλογή βεβαίως ε, στην οποία προβήκαμε ήταν πολύ ε, καλή και αυτό αφορά και την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου. Υπάρχει λοιπόν η χρηματοδοτική αυτή πτυχή για ανθρωπιστική και μη ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πρωτίστως το δημοσιονομικό σκέλος βοήθειας. Βλέπουμε ότι λαμβάνουμε, κάνουμε αποφασιστικά βήματα ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη. Ως προς τη συνιστόσα, η οποία προωθούσε μία δημοσιονομική πολιτική που ήταν αρκετά χαοτική ως προς τα Monitor Formation Centers. Θα έχουμε μία καλύτερη αλυσίδα χρηματοδότησης των διαφόρων φάσεων του εγχειρήματος λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του θέματος και τα διαφορετικά πρότυπα διαχείρισης. Σας ευχαριστώ. Όλοι μπόρεσαν να τοποθετηθούν και βεβαίως πλήθυναν τα ερωτήματα. Παρακαλώ τώρα την Επιτροπή να απαντήσει ε, στα ερωτήματα. Κύριε Τσάγκε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, κάνω κάποιες διευκρινήσεις για το τι συμβαίνει επί τόπου τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό. Στις 12 Ιανουαρίου έγινε ο σεισμός και όπως ξέρετε τα γραφεία όπου εργάζονταν η αποστολή της ΕΚΟ και όχι μόνο, όχι καταστράφηκαν, αλλά υπέσαν τέτοιες απώλειες που δεν μπορούμε πλέον να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, το προσωπικό ότι έγινε κάποια μέλη της ε, αποστολής ε, πλήγησαν αλλά εκενώθηκαν. στις 13 Ιανουαρίου η ΕΚΟ είχε ήδη κατασταθεί στο αεροδρόμιο και ήδη από ε, την ε, επόμενη μέρα, 14, οι ειδικοί πολιτικής ε, προστασίας είχαν φτάσει εκεί. Δεν υπήρξε δυσλειτουργία σε σχέση με την πρώτη αντίδραση, τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε επί τόπου. Να σε ενημερώσω για κάτι άλλο σημαντικό. Για την πρόσβαση στο Πόρτο Πράνς τρεις επιλογές έχουμε. Το λιμένα, τον αερολιμένα και το λιμάνι από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ε, οπότε χάρη στην ε, ταχεία επέμβαση των ε, ΙΠΑ που καταστάθηκε η λειτουργία στο ε, αεροδρόμιο γιατί ξέρετε ότι εδώ και δύο-τρεις ημέρες μόνο λειτουργεί ο λιμένας με περιορισμένες δυνατότητες. Ο δρόμος τώρα της ε, ήταν μη προσπελάσιμος. Ε, αυτά για να σας ε, εξηγήσω ότι ε, ούτως ή άλλως ε, επί σειρά ετών επικουρούνται οι αρχές της ΑΕΤ από τον, την επιτόπου δύναμη του ΟΗΕ. Έτσι υπάρχουν κάποιες δομές. Βέβαια ε, αποκεφαλίστηκε και πλήγει το αρχηγείο αυτής της αποστολής στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι, σε μια τέτοια καταστροφή παραδοσιακός πως η πρώτη αντίδραση έρχεται από τις τοπικές αρχές και πριν καταφτάσει η διεθνής βοήθεια ε, λειτουργεί το συστημα δυο δύο-τρει ημέρε έτσι για να υπάρχει ο ελάχιστο συντονισμό για να ξέρουμε ποιο θα φτάσει πρώτος ε, από αυτού που φέρνουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Όμω στην περίπτωση της ΑΕΤ αυτό το πρώτο κύμα τη επιτόπου αντίδραση ε, δεν υπήρχε ουσιαστικά και αυτή τη στιγμή χάνεται τρει μέρε σε μια τέτοια φυσική καταστροφή δεν γίνεται να καλύψετε αυτό το κενό. Α το έχουμε ε, κατά νου ότι ε, όχι μόνο ε, ήταν ασυνήθιστα ισχυρό ο σεισμό, αλλά και ήταν εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση επιτόπου. Ε, σε σχέση με αυτό τώρα, η τεχνογνωσία συντονισμού που είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας ε, ήδη είχε φτάσει τις πρώτες 24 ώρες. Έτσι, αυτή και μόνο η επίδοση είναι ικανοποιητική. Αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε, δείτε υπό ποιους όρους εργάζονται όλοι δίπλα στους διαδρόμους του αεροδρομίου εντάξει δεν λέω ότι υποφέρουν όπως οι σεισμόπληκτοι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργάζεται κανείς ε, με τέτοιους όρους. Για τον συντονισμό πάντοτε μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν σας πω ότι είναι τέλεια όλα ε, και υπάρχουν διάφορες πτυχέ αυτού του συντονισμού που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, ε, Συντονισμό ανάμεσα στου Ευρωπαίου και μπορώ να πω ότι λειτουργεί αισίως. Φυσικά μπορεί να αναβαθμιστεί, αλλά ήδη λειτουργεί καλά ε, και ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και ανάμεσα στις ε, διάφορες υπηρεσίες ε, της Επιτροπής. Πολιτική προστασία δηλαδή και ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, και επί που και στις Βρυξέλλες ε, αυτά τα δύο σκέλη της κατεπίουσας βοήθειας είναι σε συνεχή επικοινωνία και δεν μου έχουν επισημάνει σημαντικό εισαγωγικά επεισόδιο. Η ΜΙΚ τώρα που αναλαμβάνει το συντονισμό στις Βρυξέλλες ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, λειτουργεί ε, τέλεια και για το ανθρωπιστικό κομμάτι ο συντονισμός ανάμεσα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη ακολουθεί τη ρουτίνα. Έτσι είναι συστήματα πληροφορικής ε, που τροφοδοτούν, ε, συγγνώμη, διοικητικής που τροφοδοτούμε διαρκώς και ξέρετε είναι και μικρό το κτίριο, εν πάση περιπτώσει όλοι επικοινωνούν έτσι, τηλεφωνούν στους συναδέλφους ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέμβαση από κοινοτικό προϋπολογισμό, πολιτική προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή, έχουμε φτάσει περίπου στα 195 εκατομμύρια σήμερα. Έτσι. Αυτά, για την αυτά για τον επιτόπιο, επιτόπιο συντονισμό. Όλοι ξέρουν πόσο δύσκολο είναι και ότι η Μινουστά ε, έχει ένα κομμάτι πολιτικό και ένα κομμάτι στρατιωτικό. Ε, όλοι το ξέρουν, έτσι δεν είναι και κανένα μυστικό ότι το αστυνομικό, το στρατιωτικό κομμάτι έχει μεγαλύτερη εξουσία σε σχέση με το πολιτικό που αναλαμβάνει όμως το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και γι' αυτό το λόγο από πλευρά μα με συνεκτικό τρόπο, ε, συντονισμένο τρόπο ασκούμε πίεση ούτω ώστε το σκέλο τη ανθρωπιστική βοήθεια τη Μινουστάρε να αναδειχθεί σε σημαντικότερο κομμάτι και γίνεται σιγά σιγά έτσι, ε, για την επιτόπια παρέμβασή τους ε, και έχουν γίνει διάφορε μεταρρυθμίσει για τη λειτουργία τη ανθρωπιστική βοήθεια και βασίζονται στα κλάστερ ε, στι διάφορε ομάδε που λειτουργούν επί τόπου. Ε, ένα κλάστερ, μια ομάδα για τη στέγαση, παραδείγματο χάρη, για να προετοιμαστούν τα κέντρα στέγαση. Αν πάτε εκεί, θα εντυπωσιαστείτε από τη λεπτομέρεια, από την ακρίβεια των εργασιών συντονισμού που γίνονται επί τόπου. Ε, αυτά ε, για να ξέρετε επιχειρησιακό πόσο ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο. Τώρα, να σας μιλήσω για τις ε, αποφάσεις, τις ρυθμιστικές και για τον προϋπολογισμό. Κάθε φορά που συμβαίνει ένας σεισμός, η ώρα καταγραφής της σεισμικής δόνησης ενεργοποιεί ένα ρολόι σε σχέση με το οποίο μετράμε το χρόνο παρέμβασης. Έτσι και ε, το ποσό. 3 εκατομμύρια, σας το είπα. Χρειάζονται όμως 24 ε, ώρες. Αυτό το δημοσιονομικό εργαλείο μου επιτρέπει να ε, χρηματοδοτήσω όλες τις επιχειρήσεις ε, από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης. Δεν υπάρχει διακοπή δηλαδή. Ε, και τώρα πώς ε, λειτουργεί η υπηρεσία μας. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περνάμε μέσα από τις αρχές της ΑΕΤΙΣ για την ανθρωπιστική βοήθεια. Άμεσα συνεργαζόμαστε με τους εταίρους. Ποιοι είναι οι εταίροι μας. 186 ΜΚΟ, Ερυθρό Σταυρό, ΟΗΕ. Έχουμε συμβάσεις πλαίσιο ε, χάρη στις οποίες ε, κάνουμε άμεση εξωτερική ανάθεση. Με το που παίρνουμε την ε, απόφαση υπογράφουμε τις συμβάσεις με τις ΜΚΟ που προετοιμάζονται με το που γίνεται ο σεισμός και ξέρουν ότι ούτως ή άλλως 3 εκατομμύρια θα τα πάρουν επιτόπου και κεντρικά. Αρχίζει η επικοινωνιακή πολιτική, προετοιμάζονται να σας δώσω και ένα παράδειγμα, Πρόεδρε. Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός που είναι στη Δομινικανή ε, συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό με εμά ε, για την παροχή υποσύμου νερού Οπότε στην απόφαση τριών εκατομμυρίων είναι λογικό να πάει ένα κομμάτι στον Ερυθρό Σταυρό που άμεσα θα μετατοπιστεί, στο πάει στο Πόχτο Πχάνσε για να αρχίσει να δίνει πόσιμο νερό. Και να κάνω και ένα σχόλιο για μια παρέκκληση σε σχέση με τον δημοσιονομικό κανονισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μόλι περατώνεται ένα πρόγραμμα, η ΜΚΟ κρατάει τον εξοπλισμό έτσι, που αγόρασε για να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Ο Ερυθρό Σταυρό της Ισπανίας ε, εδώ και 10 χρόνια χρησιμοποιεί εξοπλισμό που ε, είχαν αγοράσει σε μια επιχείρηση που είχαν κάνει πριν από ε, μια δεκαετία. Για να ξέρετε ότι είναι πολύ φιδωλή έτσι, στη χρήση των πόρων η εταίροι μας. Τώρα, για τον τρόπο λειτουργίας μπορώ να δώσω κάποια επιπρόσθετα στοιχεία για τους επιπρόσθετους πόρους που ενδεχομένως χρειάζονται και για την αξιολόγηση για το UFAST και κτλ. Λοιπόν, αν είχαμε μια τέτοια δύναμη, καλό θα ήταν. Ε, δεν νομίζω ότι δυσκολεύεται κανεί να το ισχυριστεί. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί ενδεχομένω για να ληφθεί απόφαση, αλλά ταυτόχρονα οι συντονιστικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί πολιτική προστασία που έχουμε μα επιτρέπουν να καλύψουμε αυτή την απουσία τη ε, UFAST. Ε, ε, όχι ότι δεν θα ήταν χρήσιμη, αλλά δεν συνιστά αυτό και βασικό, βασική αναπηρία βασικό μειονέκτημα, έτσι, γιατί καλυπτόμαστε από το ΜΙΚ. Για τους επιπρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους, όπως σας έλεγα προηγουμένως, δεν θα σταματήσουμε τα πάντα έτσι μετά το δίμηνο. Ε, ο Στεφάν και η υπηρεσία του σίγουρα θα μας μιλήσει για τα μεσομακροπρόθεσμα, έτσι, για το πρόγραμμα Food Facility, ε, για τα τρόφιμα. Αυτό δεν αφορά κανονικά στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, μέσα σε δύο μήνες ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να υποβάλω στον Επίτροπό μου μία πρόταση παράτασης για τη χρηματοδότηση κατασκευής αντισκήνων και για την, τον εφοδιασμό σε τον επιστημιστικό εφοδιασμό. Ε, ανεφοδιασμό. Δεν μπορώ να σας πω, ε, δώσω συγκεκριμένα πόσα, θα πούνε και συναδελφοί από τον προϋπολογισμό, αλλά το πρώτο στοιχείο είναι η προσφύγη στο αποθεματικό για την κατεπίγουσα βοήθεια και τακτικά ε, και με επικοδομητικό τρόπο συνεργαζόμαστε με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ προϋπολογισμού και ευχαριστώ την Επιτροπή σας, έτσι, Ρίστο Εμπαρόδο, για την ταχύτητα με την οποία θέτε στη διάθεσή μα του πόρου που χρειαζόμαστε, οπότε ε, είναι σαφές για μένα ότι η κατεπίγουσα βοήθεια πάει στην ΑΕΤ. Εντάξει, κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι μάλλον θα χρειαστεί να προσφύγουμε σε αυτό το αποθυματικό, αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος. Ε, σε δυο τρει εβδομάδε θα έχω διαμορφώσει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για τα ποσά που ευλογοφανώ θα χρειαστούμε μέχρι το πέρας του έτους και θα συνεργαστούμε με τη ΓΔ προπολογισμού για να δώσουμε τη βέλτιστη δυνατή απάντηση. Ιδού ελπίζω να απάντησα στις βασικές ερωτήσεις σας. Α, ναι. Ε, ο κύριος Μποκρός ε, με ρώτησε κάτι για τον συντονισμό με τη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν δυσκολίες, ε, το ξέρετε. Όλοι αυθορμήτως πώς ε, δεν σπέβδουν ε, να υπαγούν στο συντονισμό του, των Ηνωμένων Εθνών, αλλά βραχυπρόθεσμα για αρρωγή προς αυτούς που είναι θαμένοι κάτω από τα ερήπια. Έχουμε το ΣΟΚ, δηλαδή ένα κέντρο επιτοπίου συντονισμού που αναλαμβάνει λοιπόν ε, τον απαιτούμενο συντονισμό για τα σωστικά ε, συνεργεία ε, για να αποσυρθούν από τα ερήπια οι πληγέντες και δεν έχω λάβει σημαντικές καταγγελίες τώρα από αυτή την πλευρά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθύντα. Ήσασταν πάρα πολύ ακριβείς στις απαντήσεις σας. Παρακαλώ. Εντάχει σας παρακαλώ γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Απλώς να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Πίτερ Ζάγκελ. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, δύο βασικά ζητήματα, η σπουδή, ο συντονισμός και τα αριθμητικά στοιχεία. Ως προς τη σπουδή της ανθρωπιστικής βοήθειας και τον άμεσο χαρακτήρα της μη ανθρωπιστικής βοήθειας αφορά την ανοικοδόμηση. Τα 100 εκατομμυρία είναι, είναι ποσό ε, διαθέσιμο άμεσα μπορεί να δαπανηθεί άμεσα. Απλώς θα πρέπει να ε, μπει σε άλλη επικεφαλίδα. Αλλά οι πληρωμές είναι έτοιμες. Και αν πληρούνται οι όροι θα δοθεί αυτό το ποσό. Η αποστολή στο τέλος της μαμάδας θα γίνει για να δούμε αν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι. Υπάρχουν και διαδικασίες ε, κατεπήγοντος άρθρα 72-73 της Συμφωνίας Κότονου ως προς τις δημόσιες προμήθειες έτσι ώστε να συνάψουμε συμβάσεις για άμεση νοικοδόμηση. Ως προς τη σπουδή δεν πρόκειται μόνο για την καταβολή πληρωμών αλλά τον μεταγενέστερο προγραμματισμό γιατί ένα από τα σφάλματά μας είναι ότι επικεντρωνόμαστε στις άμεσες ανάγκες αλλά η επίγουσα βοήθεια έχει διάρκεια δεν, μπορεί να, δεν μπορούν να αναλυφθούν οι πληρωμές από την κυβέρνηση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας χρηματοδοτικός προγραμματισμός από τώρα. Πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια, λοιπόν, υπάρχουν οι επίγουσες ε, μη ανθρωπιστικές ανάγκες. Εδώ θα δοθούν τα 100 εκατομμύρια. Ως προς το συντονισμό, μιλάμε για τα κράτη-μέλη αλλά πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία. Κινητοποιήσαμε το, την αναπτυξιακή συνιστόσα των κρατών για να έχουμε μία τάξη μεγέθους. Να δούμε ποια ποσά επαναπρογραμματίζονται και, καθώς και τους εξειδικευμένους τομείς για την οργάνωση εργασίας, έτσι ώστε να μην κάνουμε όλοι τα ίδια. Αρχίσαμε από αυτό. Θα γίνει μια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών στις 8 και στις 9 και έχουμε και την ε, άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Ανάπτυξης στις 17-18. Έχουμε έναν επιμερισμό εργασίας, τον οποίο θα αναλύσουμε. Ως προς το θέμα συντονισμού με τους άλλους φορείς, αυτό θα το προετοιμάσουμε για την διάσκεψη του Μοντρεάλ του Μαρτίου. Οι Αμερικανοί και οι Καναδοί θα συνεργαστούν μαζί μας και εδώ συνδράμουν και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα η Βραζιλία, όχι μόνο ως προς το στρατιωτικό σκέλος και η Δομινικανή Δημοκρατία καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ανοίξει τους δρόμους που τώρα είναι ανοιχτοί 24 ώρες το 24ωρο. Δεν ε, υπάρχουν πια στενοποί. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακό χάος. ώρας προς τα αριθμητικά στοιχεία για την ανοικοδόμηση είναι πολύ νωρίς να δώσουμε στοιχεία. Θα δούμε τι θα κάνει και η Παγκόσμια ε, Τράπεζα και με το ΠΝΟΥΝΤ θα γίνει μία αποστολή αξιολόγηση την επόμενη εβδομάδα. Στα πλαίσια του ΕΤΑ θα δούμε πώς θα κινηθούμε και αν χρειαστούμε επιπρόσθετες γραμμές του προπολογισμού. Δεν το ξέρω τώρα. Ως προς το Food Facility υπάρχει ένα υπόλοιπο του προγράμματος που δεν θα χρησιμοποιήσουμε για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια ε, ήταν, εντασσόταν σε ένα σχέδιο του ΦΑΟ. Ως προς την οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις ε, μελλοντικές εργασίες και μετά την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να δούμε πώς θα προβούμε στην ανοικοδόμηση του κράτους. Αλλά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Θα ήταν αυθαίρετα αυτή τη στιγμή. Το Μάρτιο νομίζω ότι θα έχουμε ε, πολλά ποσά που θα διατεθούν. Έχει σημασία να είναι πραγματικά διαθέσιμα αυτά τα ποσά μεσοπρόθεσμα, διότι μπορεί να δεσμευτεί κανείς ε, σε μία διάσκεψη και μετά να μην κάνει τίποτα. Το είδαμε πολλές φορές αυτό, άρα θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Ο Επίτροπος Ντεγκούχτ και ο Επίτροπος Πιμπάλξ ε, το τόνισαν αυτό, δηλαδή θα συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο. Όποια επιτροπή και να εμπλέκεται και να ζητά πληροφορίες θα τις έχει. Θα ενταχθεί στο σχέδιο πολιτικής υποστήριξης μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας. Ξέρουμε την IT, το πρόβλημα υπήρχε και επιτάθηκε. Άρα θα υπάρξει συνεχής διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε τους γενικούς διευθυντές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, τις παρεμβάσεις και τις απαντήσεις σας. Το Κοινοβούλιο γενικά και η Επιτροπή Προϋπολογισμών ειδικότερα θέλει να σας βοηθήσει. Έχει δεσμευθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλει να επιβραδύνει τις διαδικασίες, αντίθετα να τις επιταχύνει και αν υπάρχουν κανονισμοί που θα πρέπει να αλλάξουν για να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί θα το κάνουμε. Θα ήθελα εν παρόδο να αναφέρω τα εξή σε σχέση με τις διαδικασίες κατά πόσο είναι βραδίες ή επιταχυμένες. Θα ήθελα να πω τα εξή σε σχέση με το food facility, facility συγγνώμη, θα θέλαμε να ε, υπάρχουν χρήματα για αυτή τη συνιστόσα. Αλλά επειδή είναι μια βραδία διαδικασία θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ο πρόεδρος Μπαρόζο εδώ και δύο χρόνια είχε μία γενναιόδορη ιδέα για να βοηθήσουμε τους γεωργούς των φτωχών χωρών, ιδιαίτερα της Αφρικής, που έχουν πληγεί από την αύξηση των ε, τιμών του πετρελαίου και των σπόρων. Είχε ε, δώσει ποσά εκ των προτέρων για, την επόμενη, για τις επόμενες καλλιέργειες, για την επόμενη σπορά. Το, αυτό είχε γίνει την άνοιξη του 2008. Δηλαδή ξεπέρασε τη, τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δύο χρόνια μετά απομένουν χρήματα. Ευτυχώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι γεωργοί μπόρεσαν να σπείρουν να καλλιεργήσουν, να έχουν τη συγκομιδή τους, αλλά υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι για νεόδωρα, τα οποία επινοούμε έγκαιρα, αλλά δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προθεσμίες. Και έχετε δίκιο, κύριε Γενικέ Διευθυντά, γιατί η μεγάλη αρχηγοί και οι Ευρωπαίοι αρχηγοί, επειδή υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, ανακοινώνουν ποσά μερικές ομάδες μετά το δράμα, την τραγωδία και μετά ε, ξεχνιούνται. Εμείς, μέσα στα πλαίσια των νέων ευθυνών βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, είμαστε πληροφορημένοι εξ αρχής. Δεν θέλουμε να θέσουμε μία τροχοπέδη, αλλά να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Τσάγκελ έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτή η τραγωδία οδήγησε σε μία αυθόρμητη, ε, αυθόρμητη γενεοδορία των συμπολιτών αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε αυτά τα ποσά στα, στην ΕΚΟ ή σε άλλα ανθρωπιστικά προγράμματα ή προγράμματα διανομής τροφίμων. Αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε. Μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε το πλαίσιο προϋπολογισμού για το 2011 προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε με το σημείο 19. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ψηφοφορίες τώρα. Θα ήθελα, Ίγκε, να ασχοληθεί με το σημείο 14. Στα πλαίσια της πολιτικής κτηρίων θα θυμόσαστε ότι το Δεκέμβριο μας ζητήθηκε ένα σχέδιο ε, κτηριακής πολιτικής ε, για την Ίσπρα που είναι το κοινό κέντρο ερευνών, όπως ξέρετε, ένα από τα κοινά κέντρα ερευνών. Με βάση το άρθρο 179 του κανονισμού μας, έπρεπε να αποφασίσουμε εάν ε, επιθυμούσαμε να γνωμοθετήσουμε ή όχι. Υπό τη σύσταση της κυρίας Χολμάιερ αποφασίσαμε να γνωμοδοτήσαμε. Η κυρία Χολμάιερ ασθενεί, αλλά η κυρια χολμαιερ ασθενη αλλα η ιγκε την αντικαθιστά και θα μας προτείνει μία γνωμοδότηση. Για αν η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνη, θα αποστείλουμε μία επιστολή για την επίσημη αυτή σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ίγκε. Γκρέσλε. Έχει εξηγηθεί η κατάσταση και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τα κτίρια της Ίσπρα τα οποία εν μέρη περιέχουν αμίαντο, έχουν υποστεί και ακτινοβολία διότι ερευνητικό κέντρο ήταν. Η εισηγήτρια προτείνει συμφωνία και εγώ συμφωνώ επίσης. Σας ευχαριστώ. Είστε εκπληκτικοί σε ό,τι αφορά την νυφαλιότητα και ακρίβεια των λόγων σας. Υπόδειγμα για όλους κυρίως ε, στους ε, απογόνους των Λατίνων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγομαι. Άρα προτείνει θετική ανταπόκριση σε επιστολή. Ψήφι υπέρ της θέσεως της ηγετρίας μας για την Ίσπρα. Κατά. Αποχές. Ούτε μία αποχή. Είδω λοιπόν το αποτέλεσμα. Θα προσθέσω ότι εν ευθέτω χρόνο να δούμε αν ίσως πρέπει να στείλουμε μια αντιπροσωπεία στην Ίσπρα εκεί στις αχθές ε, της Λάγκο Ματζόρε από τα ρότερα μέρη του κόσμου όπου μπορούμε να στείλουμε ίσως και τους ε, Ιταλούς και Ιταλίδες συναδέλφους μας. Μου αρέσει η πρότασή σας για να δούμε πώς γίνεται και ε, αυτός ο παροπλισμός των πυρηνικών αντιδραστήρων ας παραμείνουμε έτσι καλοδιάθετοι και ας προχωρήσουμε στο θέμα ημεσίας διατάξεως που φέρει τον αριθμό 12 και που είναι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2010. Χρειάστηκε να συζητήσουμε με τους συντονιστές εχθές ε, το βράδυ και σήμερα το πρωί και χρειάστηκε επίσης να έλθουμε σε επαφή πάλι σήμερα το πρωί νωρίς με τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, κύριο Πιτέλα, διότι διαπιστώσαμε ότι προέκυψε πρόβλημα ερμηνείας του κανόνα αυτοπιθαρχίας για το 20% σύμφωνα με τον οποίο το Κοινοβούλιο επιβάλλει σε αυτό να μην υπερβεί στον προπολογισμό του 20% των διοικητικών δαπανών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 5 του ε, πολιετούς πλαισίου. Ε, που τηρούμε από το 1988. Στην συζήτηση επί της εκθέσεως Μάνκα για τον συμπληρωματικό αυτό είχε σημειωθεί ευρεία συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων σχετικά με το ότι η πρόταση που κάνει το Προεδρείο γίνεται δεκτή, είναι καλή, ότι χρειάζεται να μειωθεί κάπως για να παραμείνει μέσα σε αυτό το πλαφόν των 20%. Η παρουσίαση που έγινε από το Προεδρείο τότε εν καλή πίστη και επιμένω σε αυτό το καλή την πίστη όλοι μας διαθέτουμε καλή πίστη επί του προκειμένου υπήρξε κάποιο τεχνικό σφάλμα, εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες μου ή τις ευθύνες μας, περιπτώσει, για το σφάλμα αυτό. Πάντω συζητήσαμε με καλή πίστη. Ο ρόλος μου του ως Προέδρου είναι να δω να πάρουμε μια απόφαση με καλή πίστη αλλά και βεβαίω με πλήρη ενημέρωση. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις πολιτικές του ευθύνες και η ψηφοφορία της Επιτροπής Προϋπολογισμών όποιο αποτέλεσμα και να έχει θα είναι η σωστή ψηφοφορία. Πάντως, το Προεδρείο μας υπέβαλε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού και εμείς οι ίδιοι συζητήσαμε την πρόταση του εισηγητού μας θεωρώντας ότι η πρόταση του Προεδρείου που ήταν στο 20,04 της 100 ε, της κατηγορίας 5 ενώ στην πραγματικότητα μετά από διάφορες επαληθεύσεις και δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες διότι δεν μπορούμε λόγω χρόνου να ε, επισέλθουμε ψηφίσαμε έναν προϋπολογισμό αρχικό για το 2010 τον περασμένο Δεκέμβριο που ανέρχεται στο 20,2% και όχι όπως νομίζαμε 19,99. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια κατάσταση κάπως απρόσμενη που θα χρειαστεί πιθανώς να παραμείνουμε σε στενή επαφή με το Προεδρείο διότι η κατάσταση αυτή είναι νέα και για το Προεδρείο αλλά και για μας. Δεν με ανησυχεί η τελική έκφαση διότι διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρία συνένεση στην Επιτροπή Προπολογισμών για την διατήρηση των αρχικών προτάσεων του Προεδρείου. Αυτό το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι να δούμε πώς θα καταλήξουμε στη χρηματοδότηση των πρόσθετων μέτρων και πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, σύμφωνα και με την τελική απόφαση που θα ληφθεί πώς θα τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση αυτοπιθαρχίας για το πλαφόν του 20% γνωρίζοντα ότι, χωρί να το γνωρίζουμε, ήδη το έχουμε υπερβεί το πλαφόν αυτό. Αυτό είναι ο ιδιαίτερο χαρακτήρα του θέματο. Θα ζητήσω τώρα από τον εισηγητή και ευχαριστώντα τον για το έργο που κατέβαλε για το θέμα να κάνει προτάσει εις τρόπον ώστε να δούμε εάν προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία, εάν θα προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία ή εάν ο εισηγητή μα κάνει άλλη πρόταση. Πάντως ο στόχος μας είναι, και το λέω εκ των προτέρων καθαρά, είναι να δούμε ώστε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου να γίνει ψηφοφορία που θα είναι ψηφοφορία επί των προβλέψεων που μετά ε, θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την επίσημη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι ιδιαίτερη η διαδικασία αυτή και βέβαια ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα από την συνθήκη της Λισαβόνας όπου δεν υπάρχουν πλέον δύο αναγνώσεις. Υπάρχει μία ανάγνωση στην Ολομέλεια ε, για, τα, για τις προβλέψεις. Μετά πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ε, μετά προκαλεί ψηφοφορία στο ε, Συμβούλιο και επίσημη επίσης στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Εσείς, Βλαδιμίρ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να φωτίσω λίγο την κατάσταση. Τον προηγούμενο Οκτώβριο ψηφίσαμε τον προπολισμό του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με 19,87 πρώτη ανάγνωση και τελευταία γιατί είναι και δεσμευτική μετά από την έγκριση στην πρώτη αναγνώση ε, ε, ήρθαμε μετά σε συνδιαλλαγή τον Νοέμβριο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και η δική μας ε, συμμετοχή θα είναι στα 126 εκατομμύρια, δηλαδή ήρθε η κατηγορία 5 χωρίς να ανέβει ο προπολογισμό. Εφόσον όμως κατεβαίνει ε, το πλαφόν, η οροφή δηλαδή, τροποποιείται και η αναλογία. Αυτά λένε οι μαθηματικοί υπολογισμοί. Αυτό λοιπόν το 19,87 τελικώς μετά τους νέους υπολογισμούς φάνηκε να είναι 20,2%. Και αυτό ψηφίσαμε εν τέλει την προηγούμενη, την προηγούμενη χρονιά. Τα 20% της κατηγορίας 5 εμείς οι ίδιοι τα έχουμε, τα έχουμε θέσει ως στόχο το 1988. Δεν είναι νόμος, είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός του Κοινοβουλίου που επιβάλλει μια, έναν αυτοπεριορισμό σε κάποιο συγκεκριμένο όριο. Όμως δεν περιλαμβάνει τι επιπτώσεις του καθεστώτος των βουλευτών και τη συνθήκη της Λισαβόνα. Το καθεστώτος των ευρωβουλευτών φέτος οδηγεί σε αύξηση κατά 44 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν είχαμε το καθεστώς των ευρωβουλευτών ούτε την συνθήκη της Λισαβόνα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα με την οροφή. Μετά από τη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστών καταλήξαμε σε μια λύση την οποία θα σας εξηγήσω ακούσαμε όλοι, έχουμε μάλλον όλοι και δεχθεί την πρόταση του Προεδρείου για το 2010, δηλαδή να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας και είπαμε επίσης ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το, το ποσοστό του περιφερειού του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Αυτό που συζητούμε τώρα είναι να διατηρήσουμε το ποσοστό της πρώτης ανάγνωσης ώστε να έχουμε ουδέτερο προπολογισμό και μετά από τη θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνος. Πώς θα γίνει αυτό. Έχουμε τα τρία αποθεματικά. Ακίνητα, νέες προτεραιότητες και απρόσμενα γεγονότα. Στα πλαίσια αυτών των αποθεματικών θα αναζητήσουμε νέους πόρους ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τα όσα αποφασίσαμε στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό προέκυψε από ε, την συνάντηση των συντονιστών. Είναι μία πρόταση. Βεβαίω είμαι ανοιχτό και σε άλλε προτάσει. Αν κάποιο επιθυμεί να ε, κάνει άλλη πρόταση, ευχαρίστω να την ακούσω. Πολύ ωραία. Σημειώνω ότι ζητάτε το λόγο κύριε Πόρτας, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και να σχολιάσω αυτό που είπε. Για να επισπεύσω λίγο τη διαδικασία, προσπαθήσω να την επισπεύσω, έχω την εντύπωση ότι το ζήτημα τίθος εξή. εν πάση περιπτώσει θα κάνω μία πρόταση, έτσι, ε, προσθέτοντας κάτι στην παρέμβαση του εισηγητή έχουμε μια προθεσμία που πρέπει να τηρήσουμε. Έτσι, η βάση αυτών που είπαμε, η Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Νομίζω, συμφωνούμε όλοι, ότι χρειάζεται επιπρόσθετους πόρους στο Κοινοβούλιο και ότι οι προτάσεις που έκανε το Προεδρείο τη χάνουν τις αποδοχής από πλευράς ε, της πλειοψηφίας ε, των βουλευτών. Και χρειαζόμαστε τους πόρους το ταχύτερο δυνατόν. Εξού και το ενδιαφέρον του να τηρηθεί η προθεσμία του Φεβρουαρίου. Ε, πολλοί επικρίνουν για βραδίτητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βραδύτητα για την έγκριση και την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας, για την έγκριση της νέας σύνθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κρίμα θα ήταν και το Κοινοβούλιο να χάσει χρόνο εφόσον μπορεί να ασκήσει τις νέες εξουσίας του βάσει της νέας συνθήκης επειδή δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό. Οπότε ε, να τηρήσουμε την ε, προθεσμία του Φεβρουαρίου. Βέβαια, ταυτόχρονα ε, μας ευνηδιάζει αυτό το νέο στοιχείο, η σχέση ανάμεσα σε εμά και το Προεδρείο. Φυσικά θέλουμε να ε, συνεννοούμαστε με το Προεδρείο, έτσι. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων, ναι, να τη συζητάμε και να διεκπαιρεώνουμε τα ζητήματα. Αλλά δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε όταν τελικά ομονοούμε. Όπως λοιπόν ε, προτείνει ο συγητής μας και ο Γέραν Φέαρμ ε, εξάλλου παρενέβη για αυτό το θέμα στη συνεδρία των συντονιστών και ο Λάσλο, επίσημα θα πρέπει να το ξαναθίξουμε το θέμα στις σχέσεις μας με το Προεδρείο. Άρα χρειαζόμαστε μία συνεδρίαση συμφιλίωσης προτού υποβάλουμε το θέμα στην Ολομέλεια. Εξετάσαμε το χρονοδιάγραμμα. Ε, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας κανονικά θα είναι δυνατόν. 3 Φεβρουαρίου, ε, κατά πώς φαίνεται. Η πρόταση του εισηγητή μετά από πολλές συζητήσεις με όλους τους συντονιστές έγκυται στο εξή. Σήμερα θα ψηφίσουμε και θα εγκρίνουμε μια σειρά τροπολογιών που εγγράφονται στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάναμε την περασμένη φορά. Κατόπιν συνεδρίαση συμφιλίωσης για γύρω στις 3 Φεβρουαρίου με μία αντιπροσωπεία από το Προεδρείο και μία από την Κομπού και ανάλογα με την έκβαση της ε, συζήτησης αυτής ε, θα αποφασίσουμε αν χρειάζεται άλλη δική μας συνεδρίαση για να συμπληρώσουμε να τροποποιήσουμε ε, το αποτέλεσμα της σημερινής μας ψηφοφορίας. πριν την Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα, την Τρίτη ξέρω εγώ και να ψηφίσουμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Αυτή είναι η γενική ιδέα. Τώρα, αν υπάρξει ευρεία συνένεση ως προς αυτή την γραμμή, θα δούμε στις προφορικές τροπολογίες που σας έχουμε μοιράσει, που δεν σας έχουμε μοιράσει, διορθώνει ο Πρόεδρος, δύο ε, όδους μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η πρόταση του εισηγητή που αναφέρει συγκεκριμένα και υποβάλλει ψηφοφορία δύο θέματα. Πρώτον, την συμφωνία για τα νέα μέτρα που ζητά το Προεδρείο ύψους 13.400.000 ε, ευρώ. Ταυτόχρονα όμως αυτά τα 13,4 εκατομμύρια ζητά να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από κονδύλια που θα απορροφήσουμε από τα αποθεματικά. Και λεπτομερώ ε, βλέπουμε την εξοικονόμηση δαπανών ανά είδο αποθεματικού. Το πλεονέκτημα αυτή της παρουσίαση είναι η σαφήνεια και η ακρίβεια. Ε, μειονέκτημα, τα λέω δημόσια και ελεύθερα, έτσι. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Προεδρείο, θα αποφανθούμε για την εξοικονόμηση, προτού όμως να επιληφθεί του φακέλου το Προεδρείο, έχοντας ενημερωθεί για τα λάθη που έχουν γίνει ως προς την ερμηνεία. Άρα, ε, γιατί ενδέχεται να είναι έτσι η χειρή αντίδραση του Προεδρείου. Η άλλη δυνατότητα, η άλλη εναλλακτική λύση σε τι έγκυται. Με τις τροπολογίες του εισηγητή θα πούμε ότι συμφωνούμε για, τα επιπρόσθε, για τους επιπρόσθετους πόρους, 13,4 ε, εκατομμύρια, αλλά ε, δεν θα είμαστε συγκεκριμένοι σήμερα σχετικά με τη χρηματοδότηση του ποσού αυτού, αλλά θα υπερψηφίσουμε μία τροπολογία όπου η Επιτροπή Προϋπολογισμών αναθέτει εντολή σε μία αντιπροσωπεία, ώστε να έρθει σε επαφή με το Προεδρείο, ώστε να διευκρινιστούν τα απαιτούμενα μέσα για να χρηματοδοτήσουμε τα επιπρόσθετα ποσά που ζητάει το Προεδρείο με τα οποία συμφωνούμε τηρώντας όμως τους κανόνες του, του, της ε, δημοσιονομικής πειθαρχία, χωρίς όμως να αναφερθούμε σε αριθμητικά στοιχεία συγκεκριμένα. Έτσι έχουμε περιθώριο ελιγμών για να διαπραγματευτούμε με το Προεδρείο. Αυτές οι δύο ε, εκδοχές υπάρχουν. Ή θα είμαστε συγκεκριμένοι, πολύ συγκεκριμένοι, όπερ σημαίνει πως καταθέτουμε μία θέση και λέμε ότι η Επιτροπή μας επιθυμεί το, σύνολο των ε, επιπρόσθετων πόρων να χρηματοδοτηθούν από τα αποθεματικά αναφέροντας διεξοδικά πόσα κονδύλια θα πάρουμε και από ποια αποθεματικά ή δεδηλωμένα. Δίνουμε το πράσινο φως ε, στου στους πρόσθετους πόρους που ζητάει το Προεδρείο, γιατί συμφωνούμε ούτω ή άλλω. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τους ε, όρους ε, δημοσιονομικής πειθαρχία. άρρητα δηλαδή το ποσοστό του 20% και άρα να θέτουμε εντολή σε μία αντιπροσωπεία. δεν προτρέχουμε και αφήνουμε το Προεδρείο να ασκήσει την εξουσία που δικιά του είναι τελικά. Αν ναι. ε, θέσουμε πρωτατελεσμένου το Προεδρείο, δηλαδή πρέπει να βρει έναν τρόπο για να χρηματοδοτήσει τι νέε δαπάνε εξοικονομώντα από άλλε γραμμέ του προπολογισμού, ε, λοιπόν το Προεδρείο είναι αυτό που πρέπει να ε, εισηγηθεί ε, κάποια πράγματα και εμεί να τοποθετηθούμε. Ο κύριος ε, Πόρτας ε, έχει ζητήσει το λόγο, μετά ο Γιέραν, μετά η Ίγκε και μετά ο Χέλγε, η Χέλγε, συγγνώμη. Ήθελα μόνο να ενημερώσω τους συναδέλφους μου σχετικά με το ότι βγαίνω εκτός αυτή τη συμφωνίας, έτσι, που την χάνει τη αποδοχή πλειοψηφία των συντονιστών. Γιατί, πρώτον, θεωρώ ότι χρειάζεται ενίσχυση προσωπικού και στις επιτροπές και στις πολιτικές ομάδες, άρα θεωρώ ότι είναι πολιτικό σφάλμα και λειτουργικό σφάλμα να αυξήσουμε κατά 1.500 ευρώ ε, το ποσό κάθε βουλευτή για το 2010. Δεν λύνει κανένα από τα φυστάμενα προβλήματα, θα δημιουργήσει νέα προβλήματα που θα τα αντιμετωπίσουμε, θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε το 2011 και ε, τα μετέπειτα έτη. Ε, αύξηση 3.000 η αύξηση των 1.500 ευρώ. Αυτό το θέμα δεν έχει καμία συζήτηση με τη βελτίωση του διοικητικού συστήματος. Γι' αυτό είμαι κατά. Και είμαι κατά επίσης, διότι δεν μπορώ να δεχτώ την χρηματοδότηση από τα αποθεματικά. Τούτου λεχθέντος, αυτή είναι η εναλλακτική λύση που μας προτείνει ο Πρόεδρος μας. Κοιτάξτε, ε, θα πούμε συγκεκριμένα εμείς ότι θέλουμε τα 13 εκατομμύρια να χρηματοδοτηθούν από τα αποθεματικά. Οπότε τι γίνεται, 22 με 23 εκατομμύρια θα τα πάρουμε από τα αποθεματικά, αλλά στο ίδιο, ε, στο ίδιο τόπο θα τα διοχετεύσουμε. Και δεν έχουμε το θάρρος, την τόλμη, να πούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω αποφάσεις δημοσιονομικές. Δηλαδή έγινε ένα στατιστικό σφάλμα και έχουμε ένα πολιτικό στόχο από την άλλη και δεν χρειάζονται, ε, δεν μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα αποθεματικά χρειάζεται. Ένα μέτρο το οποίο δεν είναι η αύξηση κατά 1500 ευρώ του μισθού των βουλευτών. Bien, je vous remercie de la clarté. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σαφήνεια της θέσης σας. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι προτιμώ την πρόταση του εισηγητή με τα αριθμητικά στοιχεία για δύο λόγους. Καταρχήν νομίζω ότι, υπάρχει μεγάλη διαφάνεια με πού βρισκόμαστε και είμαστε πιο ευέλικτοι. Αν η συνδιαλλαγή φτάσει σε άλλο αποτέλεσμα, τότε μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογία. Δεύτερον, μας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε άλλη μια συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εάν δώσουμε αυτή την ανοιχτή εντολή, θα πρέπει να επανέλθουμε στην Επιτροπή για να αποφασίσουμε επί αριθμητικών στοιχείων. Με αυτή την ανοιχτή εντολή δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε άλλη μια συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και δεν νομίζω ότι είναι αναγκαία. Για λόγους διαφάνειας αλλά και για να αποφύγουμε μια επιπρόσθετη συνεδρίαση που δεν είναι αναγκαία θα πρέπει να δεχτούμε την πρόταση του εισηγητή με τα αριθμητικά στοιχεία που προβάλλει. Πρόεδρος. Υπό την επιφύλαξη Γκέραν ότι ενδεχομένως χρειαστούμε μια νέα συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπό αυτή την επιφύλαξη, εκτός και αν το Προεδρείο δεχτεί πλήρως τη σημερινή μας ψηφοφορία. Διαφορετικά για να τροποποιήσουμε τις ε, τροπολογίες χρειαζόμαστε μια νέα συνεδρία. Προσθέτω ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Μπορούμε να φτάσουμε και σε μια πρόταση συμβιβασμού μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα αριθμητικό στοιχείο χωρίς τις λεπτομέρειες των γραμμών όπου θέλουμε την εξοικονόμηση, την αποταμίευση αυτή. Η Ingeborg ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να ζητήσω το εξής, να μην ψηφίσουμε επί ενός εγγράφου το οποίο δεν είναι ε, έτοιμο. Ας μην το κάνουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η ψηφοφορία τώρα. Μπορούμε να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να μπούμε σε μια κατάσταση αδιεξόδου. Μας εδόθησαν δύο έγγραφα, δύο διαφορετικές προφορικές τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι οριστικό, γιατί υπάρχει, υπάρχει μεγάλο περιθώριο σφάλματος. Ο κύριος Μπόκρος. Το συζητήσαμε λεπτομερώς αυτό το θέμα σε επίπεδο συντονιστών και θα πρέπει να πω στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι δεν επετεύχθηκε ε, συμφωνία. Δεν υπήρξε συνένεση. Άρα ας μην προσπίθουμε για κάτι τέτοιο. Διαφωνώ ριζικά με κάθε διαδικασία του προϋπολογισμού που θα άρει τα αποθεματικά, διότι τα αποθεματικά είναι ύψης της σημασίας για να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας για το μέλλον. Υπ' αυτή την έννοια συμφωνώ με τον κύριο Πόρτας ο οποίος ε, είπε σαφώς ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι περικοπών δαπανών, ιδιαίτερα αυτή την αύξηση κατά 1.500 ευρώ ως προς τους ε, μισθούς για βοηθούς. Τέλος, διαφωνώ με τον Γέρεν το ζήτημα δεν είναι να αποφύγουμε μία συνεδρίαση. Αν χρειαστεί θα καθίσουμε εδώ μέρα νύχτα μέχρι ότου φτάσουμε σε μία εύλογη πρόταση. Εάν χρειαστεί συμβιβασμός θα υποστηρίξω τη δεύτερη πρόταση του Προέδρου ο οποίος είπε ας έχουμε μία ανοιχτή διαπραγμάτευση με το Προεδρείο και να δούμε ποιες νέες προτάσεις ανακύψουν και μετά να γίνει μια συνεδρίαση κομπού είτε την επόμενη εβδομάδα είτε στο Στρασβούργο και θα δούμε τι θα γίνει στο εξής. Ε, ευχαριστώ στους συναδέλφους που ήταν πολύ ακριβείς ως προς την ε, έκφραση της θέσης. του κ. Κοτμάνης. Ευχαριστώ. Δύο είναι τα ζητήματα. Μιλάμε για διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία, όπως είπαμε πριν. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε είτε να αυξήσουμε τις δαπάνες είτε όχι. Εάν δεχθούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες στον τίτλο 5, τώρα θα πρέπει να δούμε ότι κατά πόσο τα αποθεματικά στην τροπολογία 5, τα 10,4 στην κτηριακή πολιτική τα 2 εκατομμύρια και το 1 εκατομμύριο ισχύουν. Μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. τότε θα υποστηρίξω αυτή την προφορική, γιατί τι νόημα έχει να δώσουμε εντολή για συνδιαλλαγή. Μερικοί από εμά ε, θα μεταβούν, αλλά το ζήτημα είναι Τι νόημα έχει να βρεθούμε στη συνδιαλλαγή αν δεν ξέρουμε ποιοι πόροι θα διατεθούν για την αύξηση των δαπανών. Αν πάμε όμως με αυτή την πρόταση, τότε αυτά τα τρία αποθεματικά χρησιμοποιούνται για μία ε, πολιτική απόφαση. Αυτή είναι βάση συνδιαλλαγής. Αν αρχίσουμε εν λευκό στη συνδιαλλαγή και δεν αναφερθούμε στα αποθεματικά, τότε δεν θα είναι εύκολο και για τις ομάδες να λάβουν το λόγο. Υπάρχουν προτάσεις μη αύξηση δαπανών Αλλά το ζήτημα είναι να ψηφίσουμε. Θέλουμε αύξηση δαπάνω. Και τα αποθεματικά που προτείνει ο εισηγητής στη σελίδα 5, στην τροπολογία 5, σελίδα 1 ή 2, θα πρέπει να μας απασχολήσουν ως προς για το πώς, στο πώς θα κινηθούμε στο Συμβούλιο το Κοινοβούλιο. Μπορούμε να έχουμε μόνο ένα τρόπο ανάγνωσης. Εάν οι άλλοι πούν ότι αυτά τα αποθυματικά δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε, μπορούμε να βρεθούμε σε μία συνδιαλλαγή. Είναι επικίνδυνο να κινηθούμε εν λευκό. Το Προεδρείο θα πρέπει να δει από πού έρχονται αυτά τα αποθεματικά. Δηλαδή, εγώ προτείνω να υποστηρίξω με την προφορική τροπολογία C στο 5. Αλλά θα έχουμε προβλήματα με τις ε, οροφές πριν εξεύρουμε αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Καταλάβετε καλά παρακαλώ ότι εάν... Κύριε Γκοντμάνη, σε εσάς απευθύνομαι. Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ φίλε. Εάν υπερψηφίσουμε την πρόταση αναφέροντας συγκεκριμένα Ποιε είναι οι γραμμέ του προπολογισμού για τα αποθεματικά έτσι που θα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε αυτού του νέους πόρου. Δεν έχουμε πλέον τίποτα να διαπραγματευτούμε με το Προεδρείο. Τίποτα, απολύτω, ε, είναι προφανέ. αν επιθυμούμε συμφιλίω, συνδιαλλαγή με το Προεδρείο, ας αφήσουμε περιθώριο ελιγμών ε, σε αυτούς που θα αναλάβουν τη διαπραγμάτευση. Στους διαπραγματευτές πρέπει να δώσουμε ένα πλαίσιο, κάποια όρια. Για τους νέους πόρους δεχόμαστε το 13,4 από πλευράς ε, της ε, προληπτικής δράσης, ε, μάλλον της προφύλαξης έχουμε το 20% έτσι, τον δημοσιονομικό κανόνα και ανάμεσα στα δύο, καλή την πίστη θα διαπραγματευτούμε με το Προεδρείο. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη αυτή η διαπραγμάτευση παρά να πούμε ορίστε πηγαίνετε βρείτε 13,4 μάλλον να τους πούμε έχουμε 13,4 εκατομμύρια να βρούμε και θα τα πάρουμε από εκεί και μετά να πάμε να δούμε το Προεδρείο. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Ε, με απότομο τρόπο θα τοποθετηθούμε. Ε, Λάσλο. Μάλιστα, Πρόεδρε, α, ακούγοντας αυτή τη συζήτηση είναι σαφές για μένα πως δεν έχει οριμάσει ακόμη κατάσταση για να ληφθεί ε, απόφαση. Άρα επανέρχομαι στην αρχική θέση της πολιτικής μου ομάδας. αναβολή δηλαδή της απόφασης. Διαπραγμάτευση με το Προεδρείο και επαναρχόμαστε με μια πιο ισοσκελισμένη λύση. Είναι επίσης ε, σαφές ότι ομοφωνία δεν θα επιτύχουμε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, έτσι είναι η ζωή, έτσι και η πολιτική. Είναι φυσιολογικό. Αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που ε, ή θα υπάρχει πλειοψηφία που θα υιοθετήσει την πρόταση του Προεδρείου όπω ήταν, δηλαδή χάρη τη συνθήκη της Λισαβόνας και για άλλους λόγους χρειαζόμαστε αυξήσει σε κάποιες γραμμές, έτσι, αυτό το είχε προτείνει το Προεδρείο και η ε, πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Όμως, συνέπεια αυτού είναι ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα τώρα δεν μπορεί να επιληθεί, είναι σαφές. Αν δεν γίνει δεκτό και η πολιτική μου ομάδα αποκλείεται να το δεχτεί. Αν δεν δεχτεί σκεφτούμε τα ειδικά ποσά, έτσι τα συγκεκριμένα ποσά αναγραμμή για ε, απορρόφηση κονδυλίων από τα αποθαματικά. Δέχομαι αυτό που λέτε, δεν έχουμε διαπραγματευτική θέση, ζητώ συγγνώμη αγαπητέ συνάδελφε, αλλά δεν είναι σόφρον, δεν είναι τώρα. Ε, σας ε, καλώ να, να θεωρήσετε τη θέση σας. Όπως είπε και ο κύριος Μπόσκερ, Ξέρουμε που, πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα ποσά, αλλά ξέρετε την ευθύνη την έχει το Προεδρείο. Δεν θα ορίσουμε εμεί σε, σε ποιες θα υπάρξει μείωση. Αν δεχτούμε το 6 στην προφορική τροπολογία, δηλαδή εγκρίνει ε, τις εκτιμήσεις για το τροποποιητικό προϋπολογισμό σε έκτακτη συνεδρίαση, δεν χρειάζεται να περιττό να ψηφίσουμε για οποιοδήποτε ζήτημα, για ποιο λόγο θα ψηφίζαμε, πώς ακριβώς ε, θα προχωρήσουμε. Εδώ θα αποφασίσουμε για τα θέματά μας. Εδώ τα μέλη της Επιτροπής ε, δεν θα πούνε ότι όχι δεν θέλουμε έκτακτη συνεδρίαση αφού είναι έκτακτη κατάσταση συνεδρίαση της Δευτέρας δηλαδή, εντάξει δεν αρέσουν ε, στα μέλη, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνει Δευτέρα του Στρασβούργου, μπορεί να γίνει στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας. Αλλά πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να έρθουμε για να πάρουμε απόφαση. Όταν έχει βαρύτητα η κατάσταση και όταν είναι εφικτό να επιτύχουμε πλειοψηφία, να, να, ψηφίσουμε κατευθείαν, να αποφύγουμε τις συνεδρίες, αλλά δεν συμβαίνει αυτό τώρα. Οπότε, ε, καλό τα μέλη να μην ψηφίσουν. Αν ε, η πλειοψηφία ταχθεί υπέρ της ψηφοφορίας, εμείς θα καταψηφίσουμε τη λύση που λεπτομερώς αναφέρει τα ποσά και θα υπερψηφίσουμε την πρόταση για ε, διεξαγωγή έκτακτης ε, συνεδρίασης. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να επισέλθουμε τώρα σε λεπτομέρειες για το βασικό ζήτημα πέραν το ότι έχουμε μια συμφωνία έτσι, θέλουμε την αύξηση των ποσών και να χρησιμοποιηθούν οι γραμμές. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής ε, μας έχει ζητήσει το λόγο και μετά θα επανέλθω σε αυτά που είπατε. Βλαντιμίρ. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κατανοώ και τις δύο απόψεις που μόλις ακούσαμε και προτιμώ να κινηθώ πάνω στην μέση οδό. Έχω δηλαδή μια νέα πρόταση και ελπίζω να θα καταφέρουμε. Ένα πράγμα θεωρώ σημαντικό, ότι πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή για την συνδιαλλαγή, διότι χωρίς τέτοια ξεκάθαρη εντολή θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι απαιτούνται 13,4 εκατομμύρια χωρίς να πούμε, χωρίς να δηλώσουμε ακριβώς από ποια αποθεματικά θα τα αντλήσουμε. Και ας αφήσουμε μετά αυτό στο Προεδρείο, ώστε να αποφασίσει το ίδιο και να πει αυτό πού θα βρει τα κονδύλια αυτά. Αυτή είναι η πρότασή μου. Η πλειοψηφία είναι υπέρ και οι συντονιστέ στην πλειοψηφία τους τάχθηκαν υπέρ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πούμε από ποια αποθεματικά ζητούμε να προέλθουν τα χρήματα. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Ο κ. Φερνάντες. Ακούσα την τελευταία πρόταση του εισηγητού. Κύριε Πρόεδρε, Μέχρι ότου δεν έγινε επαλήθευση ότι, δεν γίνει επαλήθευση ότι υπερβήκαμε το 20% νομίζω ότι υπάρχει συνένεση ως προς την αναγκαιότητα που απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας να προβούμε σε αύξηση 13,4 εκατομμύρια για τους στόχους που ήδη ορίσαμε εκ των προτέρων. Χρειάζεται αυτή η αύξηση, αλλά τώρα η αύξηση των 1.500 ευρώ για τους βουλευτές και όχι για τους βοηθούς και τα κονδύλια για τους νέους, για το νέο προσωπικό, τους νέους υπαλλήλους και για την Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτές, αυτή η αναγκαιότητα υπάρχει. Το 20% είναι ένα, μια ενδεικτική ποσοστή αναλογία. Γιατί ένα 20% σε μια μεγάλη στήλη είναι μια, ε, μια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Σε μια μικρή στήλη δεν έχει νόημα. Γι' αυτό επιμείναμε πάντα ως προς την σταθερή αξία των δαπανών. Συμφωνώ με την θέση που προελέχθη, δηλαδή να έχουμε ε, μία σαφή εντολή διαπραγμάτευσης. Για να γίνει διαπραγμάτευση όμως δεν μπορούμε να πούμε ε, εξ αρχής πού θα γίνουν οι περικοπές. Δεν μπορούμε να πούμε εξ αρχής ε, ποια θα είναι από τα αποθεματικά που θα αγγίξουμε. Γι' αυτό συμφωνώ με τον πρόεδρο της Επιτροπής που λέει ότι θα πρέπει να δοθεί εντολή στην αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί και μπορούμε να συγκεράσουμε τις διαφορές διότι αυτή η εντολή θα πρέπει να αποσαφινιστεί και δεν είναι ασυμβίβαστη με περικοπές, ενδεχόμενες περικοπές στο αποθεματικό. Θα πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι για όσες συνεδριάσεις χρειαστούν για να επιλύσουμε αυτό το θέμα κατά τον πλέον συνενετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μη μακρηγορείτε, διότι δεν έχουμε παρά 25 ε, λεπτά ράιμερ. Ευχαριστώ. Εν ώψη της συζητήσεως που κάναμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με το Προεδρείο, κατανοώ τα επιχειρήματα των διαφόρων πλευρών. Έχουμε και είχαμε και στο παρελθόν ε, περιπτώσεις όπου το Προεδρείο έθεσε υπόψη μας πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά επεξεργασμένα και μας ευνηδίασε και αναλόγως μετά εμφανιστήκαμε εμείς ως οι καλοί ή οι κακοί της υπόθεσης αναλόγως δηλαδή με το τι στάση τηρήσαμε. Τώρα εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου αφενός μας υπέβαλαν πράγματα που ήταν σε βάση εσφαλμένων υπολογισμών, κάτι το οποίο δεν, ευθύνη, δεν βαρύνει εμάς ως ευθύνη, όλα το Προεδρείο. Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο όσον αφορά τουλάχιστον την ε, κατά συζήτηση που έγινε και την πρώτη ανάγνωση και το τι αναμένουμε μετά ως επιπτώσεις της Λισαβόνας εδώ υπάρχει μια θέση ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τα στοιχεία του διορθωτικού προπολογισμού. Δεν θέλουμε δηλαδή να ξανανοίξουμε όλα τα κουτιά ή όλα τα δοχεία. Ορισμένοι λένε, πλειοψηφία, ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τα 20% για τους λόγους. Ας μην επιτρέψουμε να προκύψει ένα τυχαίο συμπτωματικό αποτέλεσμα της ψηφοφορία που θα μας εκθέσει ως Επιτροπή Προϋπολογισμών εξετάζοντας τις διατυπώσεις που επιλέγει ο κύριος Μάνκα, ότι εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική συνεννόηση εδώ θα πρέπει να αναβάλουμε. Λέει ο Μάνκα να μειώσουμε κατά 13,4 εκατομμύρια. Ας πούμε καλύτερα μειώνοντας τα αποθεματικά ή και άλλα κονδύλια του προπολισμού κατά 13,4 εκατομμύρια. Και μια ακόμα ε, παρατήρηση κύριε Πρόεδρε, να γράψουμε μια συνοδευτική επιστολή όπου να λέμε ότι εμένουμε στο 20% και επομένως ανοίγεται η δυνατότητα εδώ το Προεδρείο να επανεγκύψει επί του θέματος και να κάνει ίσως νέες προτάσεις προσαρμογής και να μπορέσουμε τότε να προχωρήσουμε στην συνδιαλλαγή με, νέα, ε, με νέο έγγραφο του Προεδρείου. Ωραία. Χαίρομαι που μπορώ να υποφεληθώ από την σοφία του μεγάλου προκατόχου μου Μπέγκε. Μας μένουν 20 λεπτά. Όλοι έχετε ζητήσει το λόγο. Πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Εν τέλει ε, νομίζω ότι θα προκύψει ε, αποτέλεσμα της και τα πλειοψηφία. Πολλοί από εσά είπατε ότι είσαστε διατεθειμένοι να εργαστείτε και νυχθημερών, ενδεχομένω και στο Στρασβούργο. Το σημειώνω αυτό που είπατε. Και ίσω χρειαστεί να λάβετε τι ευθύνε σα. Σα κάνω την εξή πρόταση. Θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Που δεν θα έχει όμως νομικό αποτέλεσμα. Θα είναι ενδεικτική ψηφοφορία πολιτικού χαρακτήρα. Εδώ ικανοποιώ τον Λασλό. Δεν θα πούμε δηλαδή ότι εγκρίνουμε το σχέδιο προπολισμού όπως τροποποιήθηκε. Διότι είτε στερούμε σε αυτούς την δυνατότητα να διαπραγματευτούμε με το Προεδρείο, αν το πούμε αυτό, ή εάν πραγματικά προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση με το Προεδρείο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες παραχωρήσεις και άρα ενδέχεται στο τέλος, σε 15 μέρες δηλαδή, να ε, έχουμε ένα αντιφατικό αποτέλεσμα. Για λόγους διατήρησης αξιοπρέπειάς μας, ε, θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη θέση. Ψηφίζομαι, λοιπόν άνευ νομικού αποτελέσματος. Είναι όμως η ψηφοφορία μας αυτή μια πολιτική τοποθέτηση της ε, Επιτροπής Προπολογισμών, εφόσον υπάρξει βέβαια επαρκής πλειοψηφία και εγώ θέλω να επιτευχθεί μεγαλύτερη. Αν φτάσουμε σε ένα 55%-45% για ένα τέτοιο θέμα θα είναι αρκετά ε, δυσχερής η θέση μας. Πάντως, θα ήθελα να σας προτείνω μια ψηφοφορία η οποία να δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε συζήτηση και διαβούλευση με το Συμβούλιο, α, με το Προεδρείο, διορθώνει ο Πρόεδρος, και να εξηγήσουμε στο Προεδρείο ποια είναι η θέση μας, η πολιτική μας θέση δηλαδή, επί του σχεδίου που μας υπέβαλε και ε, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία που, μας, που προκύπτουν από τον νέο τρόπο υπολογισμού. με μια προφορική τροπολογία που λέει η Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκρίνει τα, τους πρόσθετους πόρους, τα πρόσθετα κονδύλια που ζητεί το Προεδρείο σε ύψος 13.400.000 ευρώ. Αυτό ήταν και η ουσία της ε, συζητήσεώς μας και ε, το περιεχόμενο της αρχικής προτάσεως του εισηγητού. Συνεχίζω. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτίθεται να χρηματοδοτήσει τα νέα αυτά μέσα με εξοικονομήσεις αντίστοιχου ύψους εντός του πλαισίου του Κοινοβουλίου του Προϋπολογισμού. Λοιπόν, θα χρηματοδοτήσει τα νέα αυτά κονδύλια από εξοικονομήσεις, από αντίστοιχου ύψου εξοικονομήσεις μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, επανερχόμαστε στην προφορική τροπολογία, σε γραπτή μορφή που το έχετε λάβει, το γάμα δηλαδή. Συνεπώς, λέει, περνώ στα αγγλικά, αποφασίζει να χορηγήσει εντολή στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών για να προχωρήσει σε συνάντηση συνδιαλλαγής με το Προεδρείο για να διευκρινιστούν τα απαραίτητα μέσα για να γίνει δεκτή η πρόταση του Προεδρείου τηρώντας όμως τους ισχύοντες κανόνες ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Δηλαδή το 20%. Βλαντιμίρ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα παρουσιάσω μια πρόταση πολύ παρόμοια με τη δική σας για να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα, αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να είναι σαφής η εντολή. Πράγμα που σημαίνει ότι κάπου πρέπει να βρούμε 13,4 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά είναι, υπάρχει και το στοιχείο του ουδέτερου του προϋπολογισμού. Είπατε ότι αν έχουμε τα τρία αυτά πράγματα, τότε είναι σαφής εντολή και μπορούμε να το ψηφίσουμε. Πρώτα, σας ευχαριστώ. Πρώτα οι συντονιστές, μετά η Γκρέσλι, ο Γιώραν. Εντάξει. Excellent. Ε, Οκ, λέει ο Γιώραν σε άψογη σφυρική. Λάσλος Σούριαν. Ε, ψηφίζουμε για την εντολή. Δεν ψηφίζουμε κανένα νομικό θέμα. Αυτό το λέω εις επίκον πάντων των παρόντων. Πρέπει να είναι λοιπόν ξεκάθαρη και εύκαμπτη η εντολή. Και μετά αυτή η φόρμουλα που προτείνει ο συγγητή, δηλαδή αυτό είναι το ποσό και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε από πού θα πρέπει να εξευρεθεί το ποσό αυτό, χωρί να λέμε αν θα είναι από αποθεματικά ή από κάποια άλλη πηγή, αυτή είναι η καλύτερη δυνατότητα που δίνουμε για τις διαπραγματεύσεις. Όλες οι λεπτομέρειες που αναγνώσατε κύριε Πρόεδρε είναι καλές, αλλά αυτή η απλουστευμένη διατύπωση είναι καλύτερη και δίνει και σε εσά ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων περισσότερες δυνατότητες να κινηθείτε. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν είμαι και εγώ σύμφωνο. Οι άλλοι συντονιστέ, η Έλγα Τρεις ώρες τα συζητάμε αυτά και από αυτά προκύπτει ότι θα αποφασίσουμε σήμερα ως πολιτικό όργανο να προχωρήσουμε σε συνδιαλλαγή με το Προεδρείο και είναι σαφές ότι πρέπει να καλύψουμε ένα κενό περίπου 13,4 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση να το πράξουμε και μετά θα χρειαστούμε μια έκτακτη συνεδρίαση και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ Έλγα. Οι φιλελεύθεροι. Λένε και αυτοί, οκ. Okay. Ε, είναι απίστευτοι, είναι απίθανοι. Και έχουν δουλέψει και όλη τη νύχτα. Η κυρία Αντρέασεν. Θα επαναλάβω τα όσα είπα στη συνάντηση των συντονιστών. Όπως και οι κύριοι Πόρτας και Βόκρος, είμαι αντίθετη με αυτή την αύξηση. Άρα για μένα δεν έχει κανένα νόημα να περιμένω οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή να αναβάλουμε. Θα καταψηφίσω ήδη σήμερα. Ο κ. Μπέγκε είπε ότι το Προεδρείο φαίνεται να λαμβάνει αποφάσεις που δεν τις έχει καλά μελετήσει. Εγώ νομίζω ότι πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Είπα και στη συνάντηση των συντονιστών ότι δεν σκεφτήκαμε τι θα γίνει εάν η απόφαση του δικαστηρίου έχει αναδρομική εφαρμογή και ζητήσει αύξηση των μισθών κατά 3,67% και αυτό θα έχει όπως είπα αναδρομική ίσχυ. Λέτε τώρα ότι θα προτείνουμε η αύξηση να καλυφθεί από εξοικονομήσεις. Εάν υπάρχουν εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό, καλύτερα να τις κρατήσουμε για να καλύψουμε την διαφορά της αύξησης των ε, μισθών. Μάλιστα, σαφής θέση. Πόρτας. Ήδη είπε ήδη ότι διαφωνείτε. Παραμένετε διαφωνών. Ναι, εσείς. Συμφωνώ με τη δική σας πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Διότι στην πρώτη τροπολογία θέλω να καταψηφίσω. Στη δεύτερη θα, θα υπερψηφίσω και στην τρίτη το ίδιο. Γιατί, τι γίνεται. Στην τρίτη Ε, να ρωτήσω και κάτι. Ε, ε, έχουμε την εντολή αλλά και τη διαπραγμάτευση για να επιστρέψουμε στο 20%, για να μην μείνουμε στο 20,2%, έτσι, γι' αυτό συμφωνώ. Très bien. Donc, monsieur est Ο κύριος Πόρτας συμφωνεί να του δώσουμε άλλο ένα λόγο για να καταψηφίσει την πρόταση. Ίγκε. Κυρία Γκρέσλε, ανησυχώ λίγο διότι όλο και περισσότερες αποφάσεις μετατίθενται από την Επιτροπή Προϋπολογισμών σε μικρότερα όργανα. Θα προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση, μετά θα προκύψουν προτάσεις και όλο αυτό γίνεται. Και έχω την εντύπωση ότι έτσι περικόπτουμε τις αρμοδιότητες ή τουλάχιστον το έργο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αντιθέτως, λέει ο Πρόεδρος, μπορούμε όντω να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία σήμερα χωρί να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι μέχρι χθε το πρωί ουδέν μέλο του Προεδρείου και ουδέν μέλο τη επιτροπή προπολογισμών, δεν γνώριζε ότι ήταν εσφαλμένα τα νούμερα. Εγώ προσπαθώ να διατηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα, να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Σέβομαι απολύτω, και αυτό είναι και το καθήκον μου, τι αρμοδιότητε παντό οργάνου του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο ήταν κακό ενημερωμένο. Έχω ανάγκη να μάθω ποια είναι η θέση του Προεδρείου όταν θα είναι καλύτερα ενημερωμένο. Η ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών ήταν αυτή ε, κακώς ενημερωμένη. Τώρα έχοντα πλήρω ενημερωθεί και γνωρίζοντας τη νέα θέση του Προεδρείου, τότε θα μπορέσει να αποφασίσει. Ε, βρίσκομαι ενώπιον αυτής αυτού του διλήμματος. Η γραμματεία τώρα βλέπουμε τον κύριο Μάνκα πως θα διαμορφωθεί ακριβώς το έγγραφο που θα υποβληθεί σε ψηφοφορία. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ε, θα ψηφίσουμε τις υπόλοιπες γραπτές τροπολογίες ε, γιατί είναι πολιτικού χαρακτήρα η ψηφοφορία. Οπότε οι νομικού χαρακτήρα τροπολογίες που θα ενταχθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα ε, ψηφίσουμε για να το υποβάλουμε συνέχεια στην Ολομέλεια θα αποσταλεί θα αναβληθεί μάλλον σε, για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά την συνδιαλλαγή με το ε, Προεδρείο. Ο εισηγητής μας χρειάζεται άλλα λίγα λεπτάκια. Monsieur le rapporteur, vous... vous... Νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει και μπορούμε να εγκρίνουμε το κείμενο υπό τους εξής όρους. Δηλαδή η προφορική τροπολογία θα αλλάξει με βάση τα όσα είπαμε σήμερα και θα δώσουμε εντολή για διαπραγματεύσεις με το Πρόεδρο. Ε, διαβάζω, διαβάζω κάπως αργά ένα μέρος στα αγγλικά, είναι στα γαλλικά. Λοιπόν, η μόνη ψηφορία που θα γίνει για αυτή την τροπολογία, έτσι, σήμερα. Δεν είναι νομικού χαρακτήρα, έτσι. είναι ένας παράγοντα παράγοντας, κάτι απρόβλεπτο και θέλουμε να το συζητήσουμε με το Προεδρείο γιατί σεβόμαστε το ρόλο του. Αν τοποθετούμαστε με οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο, θα επισύραμε την οργή του Προεδρείου, γιατί δεν θα σεβόμασταν την εξουσία του. Λοιπόν, η Επιτροπή Προπολογισμών εγκρίνει επιπρόσθετου πόρου που ζητά το Προεδρείο. Ύψου 13,4 εκατομμυρίων η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτίθεται να χρηματοδοτήσει αυτούς τους νέους πόρους με αντίστοιχη εξοικονόμηση από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Therefore, άρα, η Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει εντολή στην αντιπροσωπεία, στο κλιμάκιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών για συνεδρίαση συνδιαλλαγής με το Προεδρείο ούτως ώστε είχαμε πει clarify, specify, έτσι, να ε, διευκρινίσει ποια είναι τα απαιτούμενα ε, μέσα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Προεδρείου, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνονται με τους φυστάμενους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας με τους οποίους έχει συμφωνήσει το Κοινοβούλιο. Ωραία. Ο κύριος Πόρτας, ερώτηση διαδικαστική. Μπορούμε την πρώτη παράγραφο να την ε, ψηφίσουμε ξεχωριστά. Γιατί με τη διαδικασία εγώ συμφωνώ. Αλλά για το πολιτικό ζήτημα ζητώ χωριστή ψηφοφορία. Βεβαίω, έχετε δικαίωμα. Κύριος Χάγκλουντ. Σύντομα, Πρόεδρε, μιλήσατε για αντιπροσωπεία της Επιτροπής που θα διαπραγματευτεί. Μα ποιοι θα την ε, συναποτελούν. Οι συντονιστέ θα το αποφασίζουν ε, προφανώ, έτσι. Ε, κάθε ομάδα θα μεριμνήσει ώστε όσοι ε, έχουν ένα ειδικό βάρος, όσοι είναι νομιμοποιημένοι για αυτή τη διαδικασία, να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση, ο εισηγητή. Απλώς ήθελα να σας διαβάσω το κείμενο, γιατί υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρώτη έχει ως, όχι, ως εξής, δηλαδή 13,4 εκατομμύρια ευρώ και προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις ανάγκες με αποθεματικά και αποταμιεύσεις στο προϋπολογισμό με βάση των δύο αρχών, επί του, των δύο του προϋπολογισμού αρχών. Και το ΣΥ λέει ότι θα δώσουμε εντολή στην ε, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών για μία συνάντηση συνδιαλλαγής με το Προεδρείο έτσι ώστε να εξεύρουμε τα κατάλληλα μέσα για να αναλάβουμε τις προτάσεις του Προεδρείου τηρώντας τους κανόνες περί δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως έχουν συμφωνηθεί από το ε, Κοινοβούλιο. Εντάξει, το ίδιο μας λέτε αλλά το ανάγνωσε ο εισηγητής, αυτό είναι όλο. Ως προς την πρώτη παράγραφο που προτείνει ο εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επί της δεύτερης παραγράφου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο και λεπτό το ζήτημα και απλώς ε, νομίζω ότι διευκολύναμε τους εισηγητές, τον εισηγητή και τον πρόεδρο με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέρτμαν μου είπε ότι θέλει να θίξει ένα θέμα. Θέλετε τώρα ή στην προσεχή συνεδρίαση. Ναι, στην επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύε τη συνεδρία.